Good morning, everyone. We can make a start because all the important people are here now, except for Mrs. Gressler, of course, who will be joining us a little later, and I will chair. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ, γιατί όλοι είναι εδώ, εκτός από την κυρία Gresler, και θα προεδρεύσω εγώ μέχρι να φτάσει. Καλωσορίζω τον Επίτροπο στη συνεδρίασή μας και να ξεκινήσουμε με το σημείο 12 με την εισαγωγή από τον εκπρόσωπο του Ελεκτρικού Συνεδρίου, τον κύριο Ιτάλα. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Λοιπόν, πριν να αναφερθώ στα αποτελέσματα του ελέγχου, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το κεφάλαιο αυτό. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή των προπολογισμού της εξωτερικής δράσης ε, στη ΓΔΕΦΚΟ, ΝΙΑΡ, ΕΚΟΝ και την υπηρεσία για τα μέσα πολιτικής. Τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα είναι το μέσο για την απτυξιακή συνεργασία, το μέσο ευρωπαϊκής γειτονίας και το πρωτοεξιακό μέσο. So, for the results themselves. Για τα αποτελέσματα, το, επίπεδο, το εκτιμόμενο επίπεδο λάθος για το κεφάλαιο αυτό είναι 2,1% δηλαδή ε, λίγο πάνω από το όριο του 2%. Από 156 συναλλαγές που ελέξαμε είχαμε 24 λάθη. Σε πέντε περιπτώσεις από τις 24 η Κομισιόν είχε αρκετές πληροφορίες για να μπορέσει να προλάβει, να ανιχνεύσει και να διορθώσει τα λάθη, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες αυτές το περισσότερα από τα λάθη, 37% οφείλεται στις ελλειπείς πληροφορίες. Εδώ ο δικαιούχος ε, δεν μπορεί να αιτιολογήσει ένα ή περισσότερα τμήματα ε, του κόστους. Επίσης, ε, έχουμε γύρω στο 20% επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν δράσεις που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Για τη γάμα δέλτα νίαρ βρήκαμε αδυναμίες στην έμεση διαχείριση του προεδεξιακού μέσου, πιο συγκεκριμένα στις ε, ελεγκτικές αρχές τριών χωρών δικαιούχων. Αλβανία, Τουρκία, Σερβία. Αυτές οι αδυναμίες ε, αφορούν ε, σημαντικές ελλείψεις, οργανωτικές μεθόδους, όπως έλλειψη επαρκούς εποπτείας των αδυνομιών στην ε, κατάρτιση και την πρόσληψη του προσωπικού. Ενώ στην ε, Αλβανία και στην Σερβία οι αρχές προσπάθησαν να επιλύσουν τα λάθη που είχαν ανοιχνευτεί. Υπάρχουν σημαντικά λάθη στα τουρκικά συστήματα και φυσικά αυτό μπορεί να περιορίσει την αξιοπιστία που μπορεί να δεθεί στην Κομισιόν. Το 2016 η ΓΑΜΑ ΝΙΑΡ υλοποίησε την δεύτερη μελέτη για τα υπολοιματικά λάθη. Εμείς ε, είδαμε ότι ήταν καλό το εγχείρημα αυτό, όμως μπορεί να υπάρχει βελτίωση. Αφήθηκε ε, πολύ μεγάλη δυνατότητα κρίσης ε, στους ελεγκτές. Όμως η αιτήσια έκθεση δραστηριότητας δεν ε, κάλυψε το πεδίο εφαρμογή ε, τη μελέτη. Η μελέτη διπλού ελέγχου, διπλών λαθών, συγγνώμη, διαφέρει ε, γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί τα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο. Η μελέτη σε μερικές περιπτώσεις βασίζεται σε προηγούμενους ελέγχους και εποπτεία από άλλους ελεγκτές και δεν προβαίνει ξανά στον έλεγχο ή δεν εξετάζει λεπτομερώς τα έγγραφα εργασία. Οι μελέτες επίσης ε, απλώς χρησιμεύαν ως επισκόπηση. Τώρα, για να πάμε στα θέματα που αφορούν την υποστήριξη του προπολογισμού και τους δωρητές. Για την υποστήριξη του προπολογισμού, στήριξη του προπολογισμού, η Κομισιόν σεβάστηκε τις ε, συνθήκες πληρωμής σε συγκεκριμένα επαληθευμένα κριτήρια. Ε, ουσιαστικά εξετάζουμε τη βοήθεια που δόθηκε σε χώρες εταίρους, ε, αδυναμίες ε, σε εθνικό επίπεδο όπως διαφθορά. Αυτά οδηγούν σε λάθη στον έλεγχό μας. Η Κομισιόν έχει επαρκή ευελιξία στο να αποφασίσει αν οι γενικές συνθήκες επιλεξιμότητας γίνονται σεβαστές. Για άλλα συγκεκριμένα project, η Κομισιόν υποθέτει ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας γίνονται σεβαστοί εάν ε, το ποσό καλύπτει επαρκές επιλέξιμες δαπάνες για να καλύψει την συνεισφορά της Ένωσης. Αν όλοι οι δωρητές χρησιμοποιήσουν τις ίδιες αρχές και κριτήρια, υπάρχει κίνδυνος οι δαπάνες στο σύνολό τους να μην περιλαμβάνουν επαρκές επιλέξιμες δαπάνες για όλους τους δωρητές. Το 2016, επομένως, δεν βρήκαμε λάθη στην στήριξη των προπολογισμών ή στα project πολλαπλών δωρητών. Αν ε, ε, αποκλείσουμε ε, τα δύο αυτά από το σύνολο, έχουμε ένα εκτιμόμενο ποσοστό λαθών 2,8%. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάλεφ που τα βρήματά σας. Παρακαλώ. μικρά για τις απαντήσεις. Αξιότιμα μέλη, αξιότιμα πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριε Τσέλερ που παρουσίασε το κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις εξωτερικές μας δράσεις. Δεδομένου του πλαισίου στο οποίο ενεργούμε, χαίρομαι που τα επίπεδα σφάλματος είναι χαμηλότερα από πέρσι. Αφορά το 2,1% και έχει μειωθεί από το 2,8% το 2015 τα επίπεδα ασφάλματος ε, συστηματικά βρίσκονται κάτω από το όριο του 3% τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επίσης, ε, το εναπομείνον ποσοστό σφάλματος επίσης ε, μειώνεται κάθε χρόνο από το 3,66% το 2012 στο 1,67% το 2016. Η μελέτη για το εναπομείνον ποσοστό σφάλματος είναι βασικό μέσο για να μετρήσουμε ακριβώς τις επιδόσεις μας. Ε, μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα ε, τα τελευταία χρόνια, παρότι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να παγιώσουμε αυτές τις βελτιώσεις. Έχουμε αναλύσει διεξοδικά τα ευρήματα του ελληνικού Συνεδρίου, καθώς και τα αποτελέσματα των δικών μας μελετών για τον απομείνον ποσοστό σφάλματος και έχουμε καταλήξει στις δύο επιφυλάξεις. Η μία αφορά την διαχείριση του ε, μηχανισμού για την ειρήνη στην Αφρική. Θα επιστρέψω όταν ε, κάνω την ε, δήλωσή μου για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Παρότι το ποσοστό ενωπομείνων ποσοστό σφάλματος ήταν κάτω 2%, αποφασίσαμε να ε, ακολουθήσουμε μια προσεκτική ε, προσέγγιση και εκδώσουμε και μια διαφοροποιημένη επιφύλαξη σε σχέση με συγκεκριμένα ε, συστήματα διαχείρισης που θεωρούμε πιο επικίνδυνα, ρήψο κίνδυνα από άλλα. Ε, αυτή η επιφύλαξη θα αποτελέσει μια βάση για στοχευμένη δράση για να αντιμετωπίσουμε τι εναπομείνε αδυναμίε σε σχέση με επιχορηγήσει ε, άμεση και έμεση διαχείριση, επιχειρήσει υπό έμεση διαχείριση με διεθνεί οργανισμού και εκτιμήσει προγραμμάτων με εταιρικέ σχέσει. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ε, υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσουμε το σύστημα ελέγχου, αλλά αυτό ε, δεν αμφισβητεί τη γενική εξασφάλιση που μας παρέχει. Και τα ευρήματα του Ελληνικού Συνεδρίου και οι δικέ μα μελέτε ε, επικεντρώνονται στο κατά πόσο κάνουμε σωστά τα πράγματα. Όμω πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο κάνουμε και τα σωστά πράγματα. Το πλαίσιο αποτελεσμάτων το οποίο θεσμίσαμε το 2015 είναι ε, πολύ βασικό στοιχείο προς ε, μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα. Από το 2016 και μετά γίνονται ρητές αναφορές στα αποτελέσματα ε, στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών μηχανισμών για την χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων. Αυτό ήταν ένα κέρια σημασία βήμα για να δείξουμε την προσήλωσή μα στα αποτελέσματα προ του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Σε αυτό το πλαίσιο, ε, τα EAMR οι εκθέσεις δηλαδή ε, της ε, διαχείρισης εξωτερικής δράσης που παρουσιάζουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών είναι ε, βασικό εργαλείο διαχείρισης ε, και διαφάνους λογοδοσίας. Αυτές οι εκθέσεις παρέχουν εχέγγυα σε ό,τι αφορά τη χρηστή οικονομική διαχείριση των ε, πόρων και ταμείων μας και εντοπίζουν και συγκεκριμένα ζητήματα στις επιδόσεις μας σε ό,τι φορά μεμονωμένε επιχειρήσει. Το 2016 πετύχαμε πολύ καλού βασικού δείκτε επιδόσεων με 21 από του 24 δείκτε να ε, συνάδουν με του στόχου που είχαν τεθεί σε σχέση με 20 το 2015. Οι υπηρεσίες μου θα εξετάσουν ε, και θα τα συζητήσουν περαιτέρω αυτά τα ζητήματα μαζί σας τον Νοέμβριο. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα επί τη ευκαιρία σήμερα να υπενθυμίσω το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ενεργούμε. Ξεκινώ με το μεταναστευτικό. Πέρυσι σημειώσαμε πρόοδο στη μετανάστευση και την κινητικότητα. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Μετανάστευση, ε, το Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτη Ανάγκη για την Αφρική και η νέα εταιρική σχέση, ε, μάλλον το πλαίσιο εταιρική σχέση για την μεταναστευτική συνεργασία ήταν κέρια σημασία το 2016 για να στηρίξουμε τι ε, δεσμεύσεις, την υλοποίηση δεσμεύσεων που ελήφθησαν στη Βαλέτα. Αυτά είναι παραδείγματα των ε, προσπαθειών μας για να χειριστούμε με καλό τρόπο ε, τη μετανάστευση με σκοπό την ανάπτυξη, ενώ αντιμετωπίζουμε και τις βασικές αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης. Για πολλούς ανθρώπους η μετανάστευση είναι η μοναδική διέξοδος από τη φτώχεια. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ε, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ανάπτυξη όπου αυτά είναι πιο απαραίτητα. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο που μόλις υιοθετήθηκε θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες. Η Νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη ενδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Η εξάλληψη της φτώχειας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης παραμένει βασικός μας στόχος. Ε, θέλουμε να επενδύσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε και στην κοινή μας ασφάλεια και ευημερία. Γνωρίζουμε ότι χωρίς πραγματική ειρήνη και ασφάλεια όλα τα αναπτυξιακά ωφέλη ε, θα υπονομεύονται ε, σοβαρά και κάποιες φορές ούτε καν θα επιτυχάνονται. Γι' αυτό και αξιοποιούμε όλους τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αδυναμίες. Θέλω εδώ να είμαι σαφή. Δεν θα επικεντρωθούμε στην ειρήνη και την ασφάλεια σε βάρο των αναπτυξιακών μα στόχων, αλλά ακριβώ επειδή μα δίνουν την καλύτερη ε, δυνατότητα ε, να τους πετύχουμε πραγματικά αυτούς τους στόχους. Τέλος, πάντα, όπως πάντα λέω και σήμερα, ότι ε, η ενίσχυση των γυναικών και των κοριτσιών είναι αγρογωνία λίθος για την ανάπτυξη, ε, μία από τις ε, βασικότερες πηγές και πόρους που δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως για την βιώσιμη ανάπτυξη. Φέτος, το σχέδιο δράσης με βάση το φύλλο δείχνει ότι υπάρχει πραγματική αλλαγή πλέον, έχουμε πετύχει πραγματική αλλαγή στις νοοτροπίες και προσεγγίσεις επιτόπου, ενώ βάζουμε κατά θεμέλια για τη δράση μας τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ε, τον περασμένο μόλις μήνα ξεκινήσαμε ε, την εμβληματική και καινοτόμο ε, πρωτοβουλία Spotlight με χρηματοδότηση σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη ε, στην Γενική Συνέλευση της Νέας Υόρκης για να εξαλείψουμε την βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Αξιότιμα μέλη, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την ευημερία ε, παγκοσμίω. Με τη βοήθεια σα μπορούμε να το πάμε ακόμα καλύτερα και προσβλέπω στη συνέχιση τη συνεργασία μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτρο. Ο εισηγητής τώρα, ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση, για την απαλλαγή. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Μίμητσα και τους συνεργάτες του που είναι στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Το ελεγκτικό συνέδριο στην αρχή της συνεδρίασής μας αναφέρθηκε στα αποτελέσματα από τον έλεγχο και του τομέα αρμοδιότητος του κυρίου Χάν. Η ακρόαση έχει γίνει ήδη σχετικά στον τομέα δηλαδή βοήθεια στα πλαίσια της γειτονία δεν θα επισέλθω ούτε στη διεύρυνση, αλλά περιορίζομαι στον τομέα αρμοδιότητας του κυρίου Μίμητσα. Όμως σχετικά με τον κύριο Χάν θα υποβληθούν γραπτές ερωτήσεις γιατί έκανε κάποιες ε, επικρίσεις ε, το ελεγκτικό συνέδριο ιδιαίτερα για την έμεση διαχείριση. Γενικά χαιρετίζουμε τις θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη μείωση του ποσοστού σφάλματος. Διαπιστώνεται ότι ο προϋπολογισμός ε, δεν έχει λάθη αλλά αυτό είναι περιορισμένο όσον αφορά τη συμμόρφωση στις υποστηριζόμενες χώρες πολλές φορές υπάρχουν μεγάλα ποσοστά απάτης και διαφθοράς και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Ευχαριστούμε το ελεγκτικό συνέδριο που υπολόγισε τα σφάλματα χωρίς την στήριξη του προϋπολογισμού. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα στους ελέγχους σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων. Κάποιες ε, δαπάνες γίνονται δεκτές ενώ δεν έχουν πιστοποιηθεί. Τι μέτρα θα λάβει η Κομισιόν για να μην συμβαίνει αυτό πια στο μέλλον, αλλά να, οι πληρωμές να αναφέρονται άμεσα στη, στα παραδοτέα. Ε, τώρα, το υπολοιπόμενο είναι 67, ποσοστό λάθους, κάτω από το ε, ποσοστό σοβαρού σφάλματος ε, μειώθηκαν ε, και οι πληρωμές. Το ποσοστό σφάλματος στι πληρωμές πόσο είναι στους τομείς που κατατάσσονται ως υψηλού κινδύνου από τις γενικές διευθύνσεις, που δεν είναι και λίγοι αυτοί οι τομείς υψηλού κινδύνου. Ένα θέμα της συζήτησής μας είναι τα EAMRs. Και φέτος επαναλαμβάνω ότι η Κομισιόν με βάση το άρθρο 67 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ε, υποχρεούται να δημοσιεύει ε, τις εκθέσεις αυτές EAMR, τις εκθέσεις ε, διαχείρισης εξωτερικής δράσης. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ε, δεν μας επιτρέπει εύκολα την πρόσβαση. Πρέπει να πάμε σε έναν κλειστό χώρο περιορισμένης πρόσβασης. Θα πρέπει να περιοριστούμε στα έγγραφα που έχουμε ζητήσει και κάποιος ε, υπάλληλος εκεί πρέπει να είναι παρόν κατά την ανάγνωση των ε, εγγράφων από εμάς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η σωστή διαδικασία εν προκειμένου. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ, γιατί νομίζω ότι οι εκθέσεις αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δήλωσης αξιοπιστίας και θα πρέπει να υπάρχει ε, εμπιστοσύνη ε, από πλευρά κοινή γνώμη. Γι' αυτό χρειάζεται διαφάνεια. Πώς μπορεί να δίδεται δήλωση αξιοπιστίας, αλλά οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή να μένουν σκοτεινοί. Πήραμε τι ε, εκθέσεις ε, ήταν διαβαθμισμένα τα έγγραφα, ε, λάβαμε έγκαιρα τα έγγραφα και αυτό είναι ένα ε, βήμα μπροστά. Σε αυτά τα πλαίσια είναι ανησυχητικό το αποτέλεσμα το, του εσωτερικού ελέγχου για τα EAMR. Ο, μιλήσαμε και με τον κύριο Κράουφο, ο οποίος είναι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου και με βάση την ετήσια έκθεση του, από το και το υπηρεσιακό έγγραφο περιορίζεται στις επιδόσεις και δεν αναφέρει αν επιτεύχθησαν ή όχι οι στόχοι. Βέβαια το θέμα είναι σε ποιο βαθμό είναι αξιόπιστη μια τέτοια έκθεση. Η, κύριε Επίτροπε, οι υπηρεσίε σα τι έκαναν για να αντιμετωπιστεί αυτό το ε, πρόβλημα. Ε, εγώ δειγματοληπτικά Ε, διάβασα κάποιες εκθέσεις και πρόσεξα ότι οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίσουν διαφορετικά τις εκθέσεις. Κάποιες υπηρεσίες προχωρούν πολύ επίσημα και τυπικά, ε, άλλοι ε, μπαίνουν σε λεπτομέρειες για να εξηγήσουν γιατί δεν επιτεύχθηκαν κάποιοι στόχοι. Ένας στόχος είναι η προβληματική του φύλου στις χώρες εταίρους με τις οποίες έχουμε αναπτυξιακή συνεργασία. Θέλουμε να στηρίξουμε τη διάσταση του φύλου. Από πολλές εκθέσεις από την Αφρική και την Ασία βλέπω ότι δεν υπάρχουν πρόοδοι εδώ, διότι οι κυβερνήσεις ε, αρνούνται να συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, να δούμε αν μπορούμε και εδώ να κάνουμε κάποια πρόοδο και να έχουμε επιτυχίες. Αν δεν γίνεται μέσω της κυβέρνησης θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι διάβλοι για να δούμε πώς θα υπάρχει δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου στις χώρες αυτές. Για τις επιδόσεις, performance, η Γενική Διεύθυνση όρισε βασικούς δείκτες, γιατί ε, ο ποσοστό σφάλματος, αλλαγή κλίματος, ε, νομίζω ότι δεν είναι σωστή προσέγγιση γιατί οι δείκτες αυτοί δεν ε, δίνουν αποτελέσματα σχετικά με τις επιδόσεις. Η Γενική Διεύθυνση γιατί δεν έδωσε βασικό δείκτη για την την μετανάστευση και τους εκτοπισμούς. Ένα άλλο θέμα προσφυλές, trust funds. Οι υπηρεσίε της Κομισιόν είναι πολύ περήφανες για το Trust Fund για την Αφρική. Ε, το Κοινοβούλιο πιστεύει όμως ότι η συνεχής αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων ε, επηρεάζουν αρνητικά την διαφάνεια και τη λογοδοσία διότι ε, υπόκεινται στην δική τους διοίκηση και είναι πολλοί εκείνοι που έχουν λόγο στην εφαρμογή των στόχων. Το Κοινοβούλιο πώς μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα και να ενημερώνεται καλύτερα για τη δράση των Trust Funds για την Αφρική. Το Trust Fund για η δήλωση αξιοπιστίας δεν ε, συνοδεύτηκε από έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου της Όλαφ ή του εσωτερικού ελέγχου. Οπότε θετική δήλωση για το Trust Fund για την Αφρική που στηρίχθηκε για να δοθεί. Πέρσι το Σεπτέμβριο ο, η Κομισιόν συνολικά έκανε πρόταση κανονισμού για το Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θα δημιουργηθεί νέο μέσο δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό θεωρεί η Κομισιόν από τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Επίση, το African Peace Facility που το αναφέρατε κι εσεί το μέσο για την ειρήνη στην Αφρική, ε, μα ενδιαφέρει πολύ που βρίσκεται η συνεργασία τώρα στα πλαίσια αυτού του μέσου με την Αφρικανική Ένωση γιατί ε, εμείς είμαστε η βασική χορηγή με πάνω από 90% οπότε πρέπει να μας ενδιαφέρει αν οι στόχοι που συνοδεύουν το μέσον αυτό, ε, το χρηματοδοτικό μέσο, επιτυγχάνονται. Υπήρχε και ένα πρόγραμμα πλαίσιο, η πρώην Επίτροπος Γεωργίωβα το είχε συνάψει με την Παγκόσμια Τράπεζα. Σε ποιο βαθμό η χρηματοδότηση που συμφωνήθηκε δημιούργησε προβλήματα. Έγιναν οι πληρωμές, ε, ξεπεράστηκαν τα, το, το, το, το κατόφλι των 7% ε, που δεν επιτρέπεται με βάση το δημοσιονομικό κανονισμό και τι πιστεύετε κύριε Επίτροπε ε, για το γεγονός ότι αμείβεται η Παγκόσμια Τράπεζα για συναλλαγές που ανήκουν στις βασικές της δραστηριότητες. Ε, τώρα για την ε, Τράπεζα Επενδύσεων ε, ξέρετε ότι οι υπάλληλοι της Τράπεζας Επενδύσεων παίρνουν πόνους. Αυτό πώς επηρεάζει το κόστος διαχείρισης των trust funds. Είναι διοικητικά κόστη αυτά. Το Μπέγκου ήταν το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο, το trust fund. Και το Trust Fund για την Κολομβία, για τον Μπεγκού. Έχουμε ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, και το ευχαριστούμε γι' αυτό. Οπότε μπορούμε εκεί λεπτομερώς να συζητήσουμε. Ένα μόνιμο θέμα είναι ότι εκεί όπου δίνει βοήθεια η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει κονδύλια πρέπει να είμαστε ορατοί, συνεργαζόμεθα με πολλούς εταίρους στον τομέα αυτό και το ερώτημα είναι το εξής. Εκεί όπου είμαστε οι βασικοί χορηγοί, βασικοί χρηματοδότες, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εκείνοι που ε, παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η βοήθεια προέρχεται από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το προβάλλουν αυτό. Έκανα πολλές επισκέψεις σε χώρες όπου δραστηριοποιούμεθα και δεν ε, προβάλλεται αυτό όπως πρέπει σε ανθρωπιστικά προγράμματα στη Λιβύη, την Τουρκία, το Λίβανο και στο Ιράκ. Πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει καθόλου ποιοι πληρώνουν. Δηλαδή βλέπουν να παρέχονται υπηρεσίες από κάποιες, ε, κάποιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, αλλά Ε, δεν γνωρίζουν την ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των οργανισμών. Επίσης, ε, αξιοποίηση των trust funds. Ένα μικρότερο θέμα για τον ΦΑΟ, που δεν είναι οργάνωση της Ένωσης, ε, καλύφθηκαν, γιατί ΦΑΟ καλύφθηκαν έξοδα ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή είναι η μόνη η οποία θα πρέπει να πληρώνει τις ε, εργασίες, το επικοινωνιακό έργο της ΦΑΟ. Ευχαριστώ κυρία Τσέλερ. Είχαμε πολλές ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Ίσως ο Επίτροπος οι συνεργάτες του να μπορούσαν να απαντήσουν καταρχήν και μετά να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Τσέλερ, που είστε μέλος του Κοινοβουλίου και βουλευτή και εισηγητής. Όταν ε, συζητούμε τη συνολική επίδοση και τον έλεγχο των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική δράση και τα μέσα και των μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να τα δούμε όλα αυτά σε ένα σωστό πλαίσιο. Το συνολικό ποσοστό των λαθών μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, από τη μία χρονιά στην άλλη. Έτσι λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πολύ μικρότερο τμήμα σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο χρηματοδότησης για τα αναπτυξιακά μας έργα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποια μέσα και εργαλεία επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να συνεργαστούμε προκειμένου να πετύχουμε τον ορθό αντίκτυπο και τη σωστή χρήση των εργαλείων αυτών. για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο ποσοστό λάθους στα προγράμματα. Η έκθεση μας ε, η έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις ε, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο λογοδοσία για την Κομισιόν. Είμαι ικανοποιημένο. Επειδή δώσαμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το εργαλείο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας απαλλαγής για το 2016, αυτό όμως υπήρχε στην ε, κοινή στρατηγική εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, ε, οι κύριοι δείκτες ε, επιδόσεων παρουσιάζονται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση της ΓΑΜΑ και στέλνονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία για τις AMRs, για τις ετήσιες εκθέσεις. Έχουμε το θέμα του απορρίτου για τις AMR, των αιτήσεων εκθέσεων για τη διαχείριση. Η διαδικασία είναι όπως την περιγράψατε και κλεισμένων των θυρών. Και είναι κάτι που υλοποιείται υπό το τεκμήριο ότι κάποιος από αυτούς Κάποιοι από αυτούς τους δείκτες και κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να διατηρηθούν ε, απόρριτα. Όμως, θα θυμάστε κι εσείς, γιατί έχετε εμπειρία στο Κοινοβούλιο, όποτε οι βουλευτές ε, αναφέρονται σε κάποιες διαδικασίες ότι θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς, ή να αλλάξουν, ε, ίσως χρειάστηκε κάπως περισσότερος χρόνος για την Κομισιόν να επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως ε, εν τέλει αλλάζουμε τη διαδικασία και ερχόμαστε πολύ κοντά σε μια πραγματική διαδικασία διαφάνειας. Θα ήθελα να συνεργαστούμε λοιπόν για αυτό το θέμα, για να φτάσουμε σε τις εκθέσεις ε, για τη διαχείριση που να αντικατοπτρίζουν τη σημασία αυτού του εργαλείου. Και ένα άλλο θέμα είναι αυτό που συζητήσαμε πριν δύο χρόνια. Και αφορά την ίδια τη φύση του εργαλείου αυτό. Εδώ δεν πρόκειται περί ταυτοποίησης ε, των project που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Απλώς ε, θέλουμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις κάποια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες ε, γραμμές, ε, ας τις πούμε έτσι, σε κάποια σημεία κατά τη διάρκεια της ζωής του προγράμματος, αυτό δεν σημαίνει ότι τελικά αυτό το project θα αποτύχει. Επομένως, είναι σημαντικό να θεωρήσουμε τις ετήσιες εκθέσεις ως πραγματική ένδειξη των θεμάτων που πρέπει να επικεντρωθούμε, προκειμένου να αποφύγουμε αρνητικά αποτελέσματα. Σε σχέση με τις ε, πράξεις για τα καταδεστατηματικά ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον ε, η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τέσσερα trust fund μέχρι τώρα. Αυτά αποτελούν πρόσθετα μέσα στην ε, πιο, στα πιο παραδοσιακά αναπτυξιακά μέσα και στην εξωτερική μας δράση γενικά. Η κυρία χρήση των ε, καταπιστευματικών ταμείων ξεκίνησε από την ανάλυση των πιο αποτελεσματικών δράσεων για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της μετανάστευσης, κυρίως τα έτη 2015-2016. Αντλήσαμε το δίδαγμα ότι οι αιτίες της μετανάστευσης ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναπτυξιακές δράσεις. Προκειμένου όμως να τα καταστήσουμε αυτό αποτελεσματικό, έπρεπε να κάνουμε περισσότερα στο επίπεδο της χρηματοδότησης και ταχύτερα. Δηλαδή να περιορίσουμε το κύκλο ζωή των προγραμμάτων. Και σκεφτήκαμε ότι ένας κανονισμός, ένα μέσο καταπιστευματικού ταμείου είναι κάτι που θα μπορούσε να συνεισφέρει σε πιο στοχευμένες ταχείες δράσεις που θα πετύχαιναν πιο εύκολα το στόχο της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της χώρες προέλευσης των μεταναστών, αλλά και για να αντιμετωπιστούν κάποιες καταστάσεις κρίσης. Συμφωνώ ότι τα κατεπιστευματικά ταμεία πρέπει να την χάνουν και αυτά σοβαρού ελέγχου στο Κοινοβούλιο, αλλά να δείτε τον ίδιο το σχεδιασμό ενός Trust Fund. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή, από όταν σχεδιάστηκε το Trust Fund, ήταν παρόν, είχαμε συστάσεις, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Επιτροπών. Επίση, ε, το έχουμε συζητήσει και εδώ, σε αυτή την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αλλά και στι άλλε αρμόδιε επιτροπέ. Έχουμε και μια, αιτής, μια μηνιαία έκθεση που έρχεται από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ προϋπολογισμού και στην Επιτροπή αυτή σε σχέση με το πώς εφαρμόζουμε τον προϋπολογισμό για τα κατεπιστευματικά ταμεία. Επομένως, ε, έχουμε παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ε, σε σχέση με τις ε, συναλλαγές που αφορούν το Trust Fund. Υπάρχει βέβαια και ένα επιχείρημα ότι το Trust Fund μπορεί να κατακαιρματίσει την αναπτυξιακή βοήθεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Νομίζω ότι για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει ε, να έχουμε δράσεις οι οποίες ε, θα είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες. Θα πρέπει λοιπόν στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικού να εξετάσουμε και πώς λειτουργούν τα trust fund σε θέματα προβολής. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν ε, επισκεφτήκαμε τις ε, τοποθεσίες όπου υλοποιούνται τα προγράμματα Δηλαδή, αν πα ε, και κάπου που υλοποιείται ένα πρόγραμμα, μπορεί να μην συνειδητοποιήσει ότι αυτό το συγκεκριμένο project ε, έχει χρηματοδοτηθεί και ενίοτε εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως για κάθε project ε, είχαμε ένα τμήμα της χρηματοδότησης που αφορούσε την προβολή και την επικοινωνία. Και μαζί με τους εταίρου μας ε, που εφαρμόζουν το πρόγραμμα θέλουμε να το, υλοποιήσουμε πιο, να το χρησιμοποιήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, μαζί με τους εταίρους θέλουμε να αυξήσουμε την ε, χρήση του προϋπολογισμού προκειμένου να αυξήσουμε την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε στον κόσμο. Κοιτάξτε, μιλήσατε για κάποιες ε, κάρτες ε, ευχητήριες που στέλνονται την πρωτοχρονιά. This was also Της ΦΑΟ. Και αυτό είναι μέρος των δράσεών μας ε, για την προβολή σε συνεργασία με το ΦΑΟ. Είναι ένα παράδειγμα βέβαια που θα μπορούσε να αυξηθεί η προβολή με διάφορους τρόπους. Όπως κάναμε παραδείγματος χάρη με το φάγιο για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τις απαντήσεις. Να δώσουμε το λόγο τώρα σε άλλα μέλη. Ορισμένοι πρέπει να φύγουν σύντομα. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα αυτούς. Η Μαρτίνα, ως ασκιώδης, Πέτρη και τα Μπάρτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για τις απαντήσεις και για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Χωρισμένες ε, παρατηρήσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τον βασικό δίκτυ επίδοσης για τον απομείνον ποσοστό σφάλματος, δείχνει ε, το πραγματικό ποσοστό σφάλματος στο κλείσιμο. Ε, χαίρομαι που έχει επιτευχθεί βελτίωση από το 2012 και χαίρομαι που το 2016 βέβαια ε, το όριο αυτό είναι κάτω από το, από το επίπεδο σοβαρών ε, σφαλμάτων. Ε, αυτό που είναι σημαντικό για μένα να δω είναι η έλλειψη τεκμηρίων, το οποίο αναγνωρίστηκε ω το πιο σημαντικό σφάλμα από πλευρά του Ελληνικού Συνεδρίου. Η Επιτροπή απάντησε ότι σε πολλέ περιπτώσει η έλλειψη τεκμηρίωση οφείλεται σε λόγου ανωτέρα βία, όπω είναι η μη δυνατότητα πρόσβαση σε ε, αποδεικτικά στοιχεία εξαιτία ε, επιδημιών, σεισμών ή άλλων λόγων. Ερώτηση λοιπόν και προς την Επιτροπή και προς το Ελληνικό Συνέδριο. Μήπως θα μπορούσατε να δώσετε ε, επιπλέον ε, τεκμηρίωση για να γίνεται διάκριση σε ό,τι αφορά την ε, ανωτέρα βία σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά, για το πρόγραμμα της ε, απασχόληση των νέων που θα ξεκινήσει το 2018. Χαίρομαι που η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ θα διερευνήσει πώ μπορεί να δημιουργήσει συνέργειε σε αυτού του βασικού ε, τομεί ε, συνεργασία ε, και να εντάξει την ανική απασχόληση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά θα θέλαμε να μα ενημερώσετε γιατί πρέπει η νεολαία να λαμβάνονται υπόψη και σε άλλου τομεί όπω η μετανάστευση, επενδύσει και το καθεξή. Πώ βλέπετε εσεί αυτή τη στρατηγική. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ε, σχέδιο εξωτερικής δράσης και τα βασικά στοιχεία, πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ε, το οποίο συστάθηκε πρόσφατα, ο συμβιβασμό επετεύχθη στου τριμερείς διαλόγους τον περασμένο Ιούνιο και έχει ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο γιατί θέλει να κινητοποιήσει 44 δις ε, ευρώ επενδύσεων στην Αφρική και στην ε, ε, ευρύτερη περιφέρεια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ε, τις ε, αιτίε μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε εμείς τον αντίκτυπο και τις επιδόσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα εξετάσει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ένα έργο πώς ακριβώς πρέπει να παρουσιάζεται για να θεωρείται επιλέξιμο και από ό,τι μάθαμε δεν θα υπάρχουν ενδιαφέροντα μέρη σε αφορά την υλοποίηση του σχεδίου. Πώ θα ε, διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Ταμείο, προκειμένου να ασκεί το δικαίωμα και υποχρέωση που έχει στον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρη, θα ήθελες ε, να ρωτήσει κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Μίμητσα και τον εισηγητή κύριο Τζέλερ όπως πάντα ευχαριστούμε και ε, το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Δείξτε λίγη κατανόηση. Εδώ θα φύγω λίγο από την πεπατημένη και θα μιλήσω για την ε, δαπάνηση ε, των χρημάτων των φορολογουμένων, όπως θεωρώ εγώ θα πρέπει να γίνεται και όπως τη βλέπω εγώ. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω όμως να σταθώ στην ανάγκη για αλλαγή. Όσο μιλάμε για το, με βάση το σημερινό πλαίσιο κανόνων, δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή. Εγώ λοιπόν δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθύνω έκκληση να κάνουμε κάτι περισσότερο. Το εκτιμώ, κύριε Επίτροπο, όταν λέτε ότι γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ε, θέλει να ακολουθεί την βούληση του Κοινοβουλίου για αλλαγή. Όμως αυτό παίρνει χρόνο και θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί. Αν λάβουμε υπόψη το ιστορικό των συζητήσεων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτά τα θέματα μας έχουν απασχολήσει και τα έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό πλέον. Μία μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια που θέλω να επισημάνω. Μιλήσατε για τα EAMR και θεωρείτε, όπως είπατε, ότι είναι ε, ένα διαφανές ε, μέσο λογοδοσίας. Αυτό είναι μια μικρή μόνο υποσημείωση, μια μικρή μόνο ε, παρατήρηση του ευρύτερου πλαισίου με το οποίο εγώ διαφωνώ. Το ευρύτερο πλαίσιο τώρα, μετανάστευση. Και μετά έχουμε μια μακροσκελή περιγραφή των ε, μέτρων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Ναι, βεβαίω. Όμω τώρα θα περάσω στην ουσία της παρέμβασή μου. Ε, πρέπει να αλλάξουμε το σημείο εστίαση. Πραγματικά να το αλλάξουμε. και όλα αυτά τα λόγια που έχουμε πει εδώ και τόσα χρόνια να τα κάνουμε επιτέλους πράξη. Με άλλα λόγια, πρέπει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στα αποτελέσματα. Τι αποτελέσματα πετυχαίνουμε με τα χρήματά μας. Κατανοώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο, ε, να γίνει αυτό στον δικό σας τομέα εξωτερικής δράσης, αναπτυξιακής βοήθειας κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να μετρήσουμε κάθε φορά ε, τι απόδοση λάβαμε από το κάθε ευρώ που δαπανίσαμε. Δεν περιμένω να μου πείτε ότι για κάθε ευρώ που δαπανίσαμε πήραμε 0,80 ή 1,30. Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Όμως όλα αυτά συνδέονται με την ε, δική μας ε, στάση απέναντι στην αλλαγή και η αλλαγή θα ξεκινήσει από, ε, από εσάς ανεξάρτητα, ή από εμάς ανεξάρτητα από το που και ποιοι είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από το Ελληνικό Συνέδριο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Κοινοβούλιο και είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Όποια πλευρά και αν εκπροσωπούμε, λοιπόν, όταν παρατηρούμε ότι δαπανούμε κονδύλια μόνο και μόνο επειδή μας έχουν ε, ε, εκχωρηθεί και πρέπει να τα δαπανίσουμε, ήδη δεν πάμε καλά. Ήδη ακολουθούμε λάθος δρόμο. Ακούμε, έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές την έκφραση ότι θα επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα σε ό,τι φορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Σε αυτού του διαδρόμου θα ακούμε συνεχώς, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία τη αλλαγή. και μην ακολουθείτε, μην κολλάτε μάλλον στους κανόνες, γιατί δεν θα έρθει από εκεί η αλλαγή. Η πραγματική αλλαγή θα ξεκινήσει όταν υπερβούμε αυτούς τους κανόνες. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό, αλλιώς δεν θα πάμε πουθενά. Ιδίω όταν δεν ακολουθείτε και του ιστορικούς κανόνε. Και πρέπει να πω, κλείνοντα, ότι αυτέ οι αιτήσει εκθέσεις ε, διαχείριση εξωτερική δράση έχουν σαφείς κανόνε του οποίου έχουμε θεσπίσει και δεν ακολουθούμε. Τελικά, λοιπόν, οι πολίτε που μα παρακολουθούν δεν θα καταλάβουν εκτό και αν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία τη αλλαγή. Ευχαριστώ. Bart. Ευχαριστώ, Μπάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και το επιτελείο σας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είστε κάτω από το ε, επίπεδο του 4% στα ποσοστά σφάλματος και τώρα 2,1%. Συγχαρητήρια λοιπόν πρέπει να σας δώσω. Πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερως ε, το έργο το δικό σας και του επιτελείου σας. Στη Γενική Διεύθυνση πραγματικά γίνεται ποιοτική δουλειά και σήμερα το πρωί το αναγνώρισα αυτό στο Fair Trade Breakfast, ένα πρόγευμα το οποίο ε, διοργανώθηκε και εκεί ε, πήρε το λόγο και ο, Ροντέλφο Ρομπέρτο Ριντόλφη για τον για τον τρόπο με τον οποίο ε, υποδεθήκατε για τους ευρωβουλευτές. Πραγματικά ε, έδωσε νέα πνοή στη συζήτηση η στάση του. Ξεκινήσατε στην ομιλία σας ε, με το καταστηματικό ταμείο για την Αφρική που θέλει να καταπολεμήσει τις ε, βασικές αιτίες ε, που οδηγούν στην μετανάστευση. Είναι ένα σημαντικό ταμείο το οποίο χρηματοδοτείται από τα κονδύλια της αναπτυξιακής συνεργασίας. Όμως σημαντικό τμήμα αυτών των κονδυλίων δεν ε, προσανατολίζεται πραγματικά στην καταπολέμηση των αιτιών της μετανάστευσης, αλλά στην φύλαξη των συνόρων, στη θέσπιση ακτοφυλακών και ούτω καθεξής. Και εγώ νομίζω ότι έτσι κάπως παρεμβαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο στον προπολογισμό τη αναπτυξιακή συνεργασία. Μπορούμε να συζητήσουμε τι θα γίνει με τη φύλεξη των συνόρων, αλλά εγώ θέτω το ερώτημα γιατί αυτό να καλυφθεί από τα χρήματα τη αναπτυξιακή συνεργασία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όλα αυτά τα δις που δαπανώνται στο καταπιστευματικό ταμείο στην Αφρική, από αυτά τα χρήματα πόσα θα πάνε πραγματικά στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην εξάλληψη των βασικών αιτιών της μετανάστευσης και πόσα χρήματα θα πάνε στη μετανάστευση. Διάβασα πρόσφατα ότι 35 εκατομμύρια θα πάνε ε, στο ε, στην ναυτική δύναμη της ε, Αιγύπτου για την ε, δημιουργία της ε, ακτοφυλακής. 35 εκατομμύρια τώρα για τέτοια πράγματα δεν νομίζω ότι πρέπει να έρχονται από αυτό τον κορβανά. Ναι, τα είπατε ότι πρέπει πραγματικά κάτι να κάνουμε για την Αφρική, να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή μας συνεργασία, την στήριξή μας, όχι μόνο με κονδύλια αλλά και με έργα, ε, να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτή την πολιτική, αλλά μήπω θα έπρεπε να τα κοιτάξουμε τα πράγματα λίγο ευρύτερα, κύριε Επίτροπε. κάνατε πολύ σημαντική και χρήσιμη δουλειά που σίγουρα συμβάλλει στην κατάρτιση πολλών ανθρώπων. Όντως πολλοί άνθρωποι στην Αφρική ε, έχουν και πάλι προοπτική για το μέλλον, εξαιρετικά. Αλλά πού είναι η συνέπεια της ευρωπαϊκής πολιτικής στο σύνολό τη. Έχουμε μια εμπορική πολιτική που πολύ συχνά σφάλει. Έχουμε μια γεωργική πολιτική, πολιτική αλληλείας που επιδρά αρνητικά στο μέλλον των Αφρικανών πολιτών. Χθε έδωσε το παράδειγμα στον Επίτροπο Έτιγκερ σε ό,τι αφορά την γεωργική πολιτική που έχουμε καταργήσει τις ποσοστώσεις ε, στο γάλα ε, και έτσι δημιουργείται σκόνη γάλακτος η οποία ε, αποθηκεύεται και μέσω της εμπορικής μας πολιτικής ουσιαστικά κάνουμε ένα dumping, ξεφορτωνόμαστε αυτή την, αυτό το προϊόν στις αφρικανικές αγορές. Για παράδειγμα, στην Ιγυρία η τιμή του γάλακτος είναι 800 με 900 ε, CFVA αναλύτρο το τοπικό νόμισμα για το γάλα που παράγεται εκεί. Ενώ το γάλα που πωλείται εκεί και προέρχεται από τη δική μας σκόνη γάλακτος είναι 300 CVA, το 1 τρίτο. Μα πώς γίνεται μετά να απορούμε ε, που δεν ε, έχουν μέλλον οι Αφρικανοί γεωργοί όταν η τιμή του δικού τους γάλακτος είναι τριπλάσια. Όταν αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν την Ήπεθρο και πάνε στην πόλη. Έτσι είπατε κι εσείς ότι δεν έχουν μέλλον, φεύγουν από την Ήπεθρο, πάνε στις πόλεις. Και αν δεν βρίσκουν και εκεί μέλλον, ε, τότε προσπαθούν να πάνε στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για το γάλα, το ίδιο ισχύει και για τα κοτόπουλα και τα προϊόντα πουλερικών που ε, εξάγουμε προς την Αφρική. Πρόσφατα διάβασα ότι από τους ε, στόλους, ε, τους αλληλευτικούς που έχουμε, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, πάνε στην Νιγηρία και στη Μαυριτανία και έτσι δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στους Αφρικανούς αλληλείς. Επομένως, κύριε Επίτροπε, Μπορούμε να επενδύσουμε πολλά για την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά τελικά πού είναι η συνοχή σε αυτή την πολιτική που έχουμε της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ ε, του Επιτρόπου Αλληλείας, Γεωργίας και ούτω καθεξής για να επισημάνατε τα κακοσκήμενα Και εσείς με τη δική σας πολιτική ε, επιστρέφετε κάτι στους Αφρικανούς, παρέχετε κάτι τελικά. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί στο τραπέζι όταν εξετάζουμε την σωστή δαπάνηση των κονδυλίων μας. Ευχαριστώ. Next speaker, Mr. Salafranca. Ευχαριστώ, κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε εδώ για να αναλύσουμε με τον Επίτροπο και με τις υπηρεσίες του την απαλλαγή του 2016 και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία για θέματα με τα οποία δεν συμφωνούμε σε σχέση με τις πολιτικές να τα θέσουμε σε άλλους επιτρόπους. Εγώ νομίζω ότι τώρα βλέπουμε μια βελτίωση στο ποσοστό λάθος και όλοι πρέπει να χαιρόμαστε για αυτή τη θετική εξέλιξη. Επίσης πιστεύω, και το εξήγησε και ο κύριος Σαβάρμα, ότι εδώ δεν θέλουμε μόνο να μειώσουμε τα ποσοστά λάθους, αλλά θέλουμε και αναπτυξιακές ε, πολιτικές να πετύχουν τους προβλεπόμενους στόχους. Νομίζω ότι αυτό είναι μια λογική και δυναμική που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε και για μελλοντικέ εξελίξεις. Εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Επίτροπο πριν να αποχωρήσω Λυπάμαι κύριε πίτροπε, πρέπει να φύγω γρήγορα για μια ψηφοφορία. Μου φαίνεται όμως ε, σημαντικό να πω το εξή. Ε, δεδομένων των ε, πρόσθετων ευθυνών που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομεί που εμπίπτουν στη δική σας αρμοδιότητα και υπάρχει ιδιαίτερα πολύπλοκη χρηματοοικονομική και δημοσιονομική διαχείριση σε ποιο βαθμό μπορείτε εσείς και φυσικά όλοι γνωρίζουμε τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός ως προς τους ανθρώπινους πόρους, σε ποιο βαθμό εσείς έχετε αύξηση μέσων για να αντιμετωπίσετε κάποια καθήκοντα που πρέπει να αναλάβετε. Και φυσικά σκέφτομαι ένα θέμα που συζητήθηκε σήμερα το πρωί και αποτελεί μέρος των παρατηρήσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου, έχει να κάνει με τις ε, βοήθειες ε, για να καταπολεμήσουμε τις ε, συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι εσείς δεν μπορούσατε να αποκτήσετε πρόσθετους ανθρώπινους πόρους για να διαχειριστείτε πολύ μεγάλα ποσά. Λυπάμαι που δεν μπορώ να μείνω για να ακούσω την απάντησή σας, όμως είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να ζητάμε και θαύματα για την οικονομική διαχείριση αν δεν υπάρχουν και απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι. Και εγώ πιστεύω ότι ακριβώς σε αυτό το θέμα της μετανάστευσης το άχθος είναι πάρα πολύ μεγάλο και η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει και τα επαρκή μέσα για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα καθήκοντα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, κάποιοι συνάδελφοι πρέπει να φύγουν κύριε Επίτροπε, αλλά ίσως τώρα θα μπορούσαμε να σας δώσουμε το λόγο για να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Και τις προτάσεις σε σχέση με την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε Πολύ σύντομα ξαναγυρίζω στους βασικούς δείκτες επιδόσεων και στις εκθέσεις της εξωτερικής δράσης για τη διαχείριση. Θυμίζω ότι το Νοέμβριο τα κλιμάκια από την Γενική Διεύθυνση Ντεύκο και ΝΙΕΡ θα έρθουν εδώ στην Επιτροπή σας και θα αναφέρουν όλες τις λεπτομέρειες που ενδεχομένως θα αποτελέσουν τη συνολική προσέγγιση στα EAMR, στις εκθέσεις αυτές, για να είναι αποτελεσματικό μέσον που θα μας επιτρέψει να έχουμε συνεχή παρακολούθηση και να εξασφαλίζουμε λογοδοσία. Θα είναι ένα μέσον, ένα εργαλείο λογοδοσίας καθ' όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων. Τώρα, για το καταπιστευματικό ταμείο. Προτείνω να οργανώσουμε μια συζήτηση θεματική, όπου θα εξετάσουμε τα trust funds και θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να συμβάλλουν στο παρόν μείγμα της αναπτυξιακής συνεργασίας, του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας. Και σε ποιο βαθμό αξίζει να έχουμε ένα μέσον ταχείας ε, υλοποίησης. Γιατί πολλές φορές μέχρι τώρα συμμετείχαμε στα trust funds άλλων και ε, ε, ε, πληρώναμε στα συστήματα της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του, του Δεν είχαμε δικά μας τέτοια trust funds. Ας καθίσουμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αξιοποιηθούν ιδιαίτερα στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Οι περισσότερες ερωτήσεις και προτάσεις των κυρίων βουλευτών θα πρέπει να περάσουν στο πλαίσιο της συζήτησης για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλήσαμε επίσης και για κάποιες πτυχές των ποσοστών σφαλμάτων. Ένα θέμα είναι η έλλειψη τεκμηρίωσης. Πρέπει και πάλι εδώ να έχουμε υπόψη μας ότι η, όλη η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και τα χρηματοδοτικά μέσα λαμβάνουν χώρα σε πολύ επικίνδυνα και απρόβλεπτα πολλές φορές περιβάλλοντα στις χώρες εταίρους όλο τον κόσμο. Οπότε η έλλειψη σωστής τεκμηρίωσης και μιας βάσης δεδομένων ε, δεν ε, είναι ίδια όπως όταν χρηματοδοτούμε ας πούμε από τον προϋπολογισμό μας γεωργικά ε, προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνοχή, το Γεωργικό Ταμείο και από την άλλη έχω, ή αν έχουμε αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ε, Ήμπισα ή κάπου αλλού στον κόσμο. Αλλά όπως ε, ε, είπε και ο αξιότιμος βουλευτής, ότι θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπες διαδικασίες, στάνταρ διαδικασίες, που θα επιτρέπουν την τεκμηρίωση ή θα ε, μειώνουν την έλλειψη τεκμηρίωσης σε μεγάλο βαθμό. Στο νέο Ευρωπαϊκό Κονσένσους για την Ανάπτυξη θεωρούμε ότι η αναπτυξιακή συνεργασία προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μία ε, διάσταση γενικότερη που επιτρέπει την υλοποίηση όχι μόνο ενός στόχου μεμονωμένου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ε, εντάσσει την νεολαία, τα, τα έργα για την νεολαία, για την ανάπτυξη, για την απασχόληση και αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφή στο Νοέμβριο στο Αμπιτζάν, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική ε, Ένωση. Αυτή θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις για τους νέους. Αυτή τη φορά θα είναι στην Αφρική. Ε, αλλά όλα τα αναπτυξιακά έργα θα πρέπει να συμβάλλουν συγκεκριμένα και στην ένταξη των νέων στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στη χώρα τους. Αρχίσαμε τώρα, ε, θέσαμε σε εφαρμογή και ένα άλλο μέσον, ε, σχέδιο, σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα χρησιμοποιήσουμε αυτές, αυτά τα μέσα συνδυάζοντας επενδύσεις από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και θα δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσεις. Είναι σημαντικό το νέο αυτό χρηματοδοτικό μέσο να μπορεί να μετράει τον αντίκτυπο, δηλαδή σε ποιο βαθμό συμβάλλει στην εκρίζωση των ε, αιτίων της, μεταφράσης, μετανάστευσης που και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες εταίρους. Το πλαίσιο των αποτελεσμάτων που αναπτύξαμε είναι μεγάλο βήμα μπροστά. Δεν πρέπει να μετράμε. Πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε τα χρήματα που βάζουμε στην αναπτυξιακή συνεργασία. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα την απόδοση όλων που έχουν όλα αυτά. Δεν πρέπει να κολλάμε δηλαδή στα νούμερα των χρηματικών ποσών, αλλά στον αριθμό των ανθρώπων που ωφελούνται από τα έργα μας. Το 2015, πως αργά, ε, αρχίσαμε να ακολουθούμε αυτό το πλαίσιο που βασίζεται στα αποτελέσματα και τώρα το έχουμε συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση. Ε, είναι αυτή μια πρώτη μπροσούρα ενημερωτικό ε, φυλάδιο όπου αναφέρομαι τους άμεσα ωφεληθέντες από τα προγράμματα. Γιατί αν πούμε επενδύσαμε δύο δις σε κάποια προγράμματα, κανείς δεν θα καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Ιδιαίτερα οι εταίρες στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν προσλαμβάνουσα τι είναι ένα δις και τι μπορεί να επιτύχει. Αν όμως πείτε ότι ένα εκατομμύριο χιλιάδες άνθρωποι ωφελήθηκαν άμεσα από προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων την διατροφή ή 35 εκατομμύρια παιδιά και παραπάνω συμμετείχαν σε προγράμματα ε, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι πολύ καλό, ενημερωτικό. Η εστίαση στα αποτελέσματα είναι το επόμενο βήμα που θέλουμε να ε, κάνουμε. Τώρα, η διάσταση της μετανάστευσης της ε, λειτουργίας των ε, trust funds. Είπατε ότι κάποια trust fund πληρώνουν για φύλαξη συνόρων, για να εμποδίσουν κάποιον να περάσει σε άλλη χώρα ή σε μια, χώρα, σε μια άλλη χώρα. Αν δούμε την πραγματική φύση αυτών των προγραμμάτων, των trust funds, δεν είναι για να χρηματοδοτεί ε, φύλαξη, συνοριοφυλακές ή εξοπλισμό στρατιωτικό ή εξοπλισμό που θα επιτρέψει στις χώρες εταίρους να ελέγχουν τα σύνορά τους καλύτερα. Πρόκειται για τη διαχείριση των σύνορων, εκπαίδευση διευκόλυνση της γενικότερης διαχείρισης των συνόρων που ε, αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια στις χώρες εταίρους μας. Όποτε λοιπόν ε, προχωράμε σε project που αφορούν τη μετανάστευση, που είναι αναπτυξιακά, και αφορούν την παράτυπη μετανάστευση στις χώρες προέλευσης, στη ρίζα τους, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ε, διοχετεύω με τα αναπτυξιακά κονδύλια στην παρεμπόδιση της μετανάστευσης. Τι σημαίνει ε, μείωση της φτώχειας, σημαίνει και μετριασμός των μεταναστευτικών ροών και ο αναπτυξιακός αντίκτυπος ε, επηρεάζει και μειώνει τη μετανάστευση. Είναι σημαντική αυτή η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ε, ανάπτυξης σε όλα μας τα αναπτυξιακά έργα. Τώρα, η Συμφωνία Οικονομικής ε, Εταιρικής Σχέσης για και η καλύτερη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη. Πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική μας ε, συνοχής για την ανάπτυξη. Ε, όλες οι πολιτικές μας έχουν σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους ε, στις χώρες μας. Το εμπόριο είναι ένας τέτοιος στόχος. Έχουμε ένα πλαίσιο ή δημιουργούμε ένα πλαίσιο συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού στην Αφρική Ειρηνική και Καραϊβική Αλλά αν θέλετε έχουμε μια προσέγγιση αντίστροφων προτεραιοτήτων με τις συμφωνίες αυτές. Ή, για να το πω έτσι, οι συμφωνίες θεωρείται ότι ασχολούνται με θέματα ελεύθερου εμπορίου ή ελευθέρων συναλλαγών ή τασμών. Αλλά η, ιδέα είναι ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πρωτίστως πρέπει να συμβάλλουν σε καλύτερο τομέα παραγωγής, καλύτερες αλυσίδες αξίας στις χώρες εταίρους, ώστε να μπορέσουν και εκείνες να έχουν μεγαλύτερης αξίας προϊόντα που θα είναι εμπορεύσιμα. Οι συμφωνίες αυτές είναι ένα εργαλείο για να βελτιωθεί η περιφερειακή και οικονομική ολοκλήρωση και η πολιτική ολοκλήρωση. Ε, στις διάφορες χώρες της Αφρικής, ε, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής. Και μόνο όταν επιτύχουμε αυτούς τους στόχους θα έχουμε ένα αποτελεσματικό εμπορικό καθεστώς ε, και ελεύθερες συναλλαγές και μία εφαρμογή δασμών στις εισαγωγές, εξαγωγές μεταξύ μας. Το δίκαιο εμπόριο είναι σημαντικό εδώ. Το εμπόριο είναι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει, πρέπει να μπει σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την, να περάσει μέσα από την βιομηχανοποίηση, τη σωστή παραγωγή και την ε, αξιακή αλυσίδα που θα έχει ε, μεγαλύτερη αξία. Τώρα, συνολικά η, φύλαξη, διαχείριση των συνόρων και η σχέση ανάπτυξης, μετανάστευσης, ε, ε, ειρήνης και ασφάλειας. Αν δείτε όλα τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά μέσα και αυτά για την ειρήνη και την ασφάλεια, σήμερα το 96% όλης της αναπτυξιακής μας χρηματοδότησης αναφέρεται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, το 96% όλων των χρηματοδοτικών μέσων, που είναι γνήσια αναπτυξιακά μέσα. Θέλουμε να ε, αυξήσουμε αυτό το ποσοστό, αλλά σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για εκτροπή, αν θέλετε, αναπτυξιακών κονδυλίων για άλλους σκοπούς αλλιώς, αλλά αυτό το ποσοστό δεν θα ήταν τόσο υψηλό Στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να εξυγχρονίσουμε τα μέσα μας, να το κάνουμε μια σχετική συζήτηση. Σήμερα έχουμε 66 δις ανθρωπιστικής βοήθειας, ελευθερία, ανάπτυξη και 30 δις στο Ταμείο Ανάπτυξης και 17 διαφορετικά κατακαιρματισμένα χρηματοδοτικά μέσα. Οπότε μπορούμε να ε, βελτιώσουμε τη λειτουργία τους, να τροποποιήσουμε τον αριθμό των χρηματοδοτικών μέσων και να βελτιώσουμε την συνολική μας χρηματοδοτική ικανότητα. Τέλος, για τους ανθρώπινους πόρους, πάλι 66 και 30, 90, 96 δις ε, για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν λειτουργούμε σαν αναπτυξιακός οργανισμός. Πρέπει να κάνουμε εταιρικές σχέσεις με άλλους. Εδώ, στα κεντρικά μας, στις Βρυξέλλες και στις αντιπροσωπείες μας στο εξωτερικό, εργάζονται αρκετοί συνάδελφοι στον τομέα της διαχείρισης των ε, δημοσιονομικών μέσων για την ανάπτυξη. Ο αριθμός αυτός μειώνεται όμως. Ενώ εμείς θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του προσωπικού μας, των πόρων μας και δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν να ε, ότι μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό του προσωπικού που ασχολείται με την υλοποίηση των έργων. σε όλο αυτό το τεράστιο αριθμό μέσων που έχουμε για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε για τις λεπτομερείς απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ίσως ε, τώρα να ξαναδώσω το λόγο στο λεκτικό συνέδριο. Τελευταίο θα δώσω το λόγο σε εσάς κύριε Τζέλερ για να ολοκληρώσετε το λεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Οι περισσότερες ερωτήσεις απαντήθηκαν. Όμως θέλω να πω το εξής. Ουσιαστικά μέσω των ε, ερωτήσεων ε, ζητήθηκε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον προπολογισμό. Αυτό ζητά ούτω ή άλλω και το ελεκτικό συνέδριο τόσα χρόνια. Επομένω, είναι σημαντικό να το βλέπουμε και από την σκοπιά του Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σα ε, σε αυτά τα κεφάλαια. Ο κύριο Τσέλερ. Thank Derek. Und Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για τις απαντήσεις του. Πολλά θέματα που αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, πέφτουν σε βίκο αότα εδώ στο Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για την μελλοντική διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι θετικό πρέπει να λάβετε υπόψη σας ε, το γεγονός ότι ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις. Είναι θετικό διότι τα θέματα της ανάπτυξης, αναπτυξιακής συνεργασίας, αναπτυξιακής πολιτικής θεωρούνται ως ε, πολύ σημαντικός τομέας της πολιτικής. Στο παρελθόν στη Γερμανία, για παράδειγμα, όταν ε, έπρεπε να βολέψω κάποιο κομματικό στέλεχος, του ανέθεταν, του ανέθεταν την αναπτυξιακή πολιτική. Τώρα η σημασία της έχει αναβαθμιστεί και επηρεάζει πάρα πολύ, όλο και περισσότερο, και το δικό μας το μέλλον. Οπότε η στενότερη συνεργασία με την Αφρική, Ασία, Μέση Ανατολή είναι σημαντική. το Κοινοβούλιο θα είναι στο πλευρό σας νομίζω. Το θέμα των trust funds και το συγκερασμό των ε, μέσων, το αναφέρατε, την καλύτερη προβολή το είπατε. Ε, χρειάζεται ευελιξία, δεν είναι κακή ιδέα. Κάποια χρήματα από μακροπρόθεσμα έργα όπου, που δεν χρειάζονται εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού για να αντιδρούμε άμεσα σε μια καινούργια ανάγκη και να εστιάζουμε σε ένα στόχο. Ε, τα trust funds θα έπρεπε να πάρουν όμως και πρόσθετα κονδύλια από νέους δωρητές, όχι μόνο από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τα τρία-τέσσερα κράτη-μέλη που ε, ήταν έτοιμα να δώσουν χρήματα έπρεπε να βρεθούν κι άλλοι να, να, να συμβάλλουν. Και υπάρχει πολύ περιθώριο εδώ, γιατί δεν ε, ε, υπήρχε ανταπόκριση στις ε, δημοσιονομικές απαιτήσεις που διατυπώθηκαν σε σχέση με αυτά τα trust fund. Και η διοίκηση πολύ συχνά συμβαίνει να χάνει, να, οι διοικήσεις να χάνουν τον πραγματικό στόχο. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί εδώ. Για τις αιτήσιες εκθέσεις ε, δραστηριοτήτων, είναι, αυτές είναι σημαντικές για να μετράμε τις ε, επιδόσεις, τα αποτελέσματα. Σε πολλές εκθέσεις ε, αναφέρεται ότι στις αντιπροσωπείες της Ένωσης δεν υπάρχει αρκετό εκπαιδευμένο προσωπικό ούτως ώστε να, ελέγχουν τα έργα ε, στον τομέα της ανάπτυξης. Αυτό ισχύει εκεί όπου χορηγούμε ε, δημοσιονομική στήριξη. Όλες οι δαπάνες ε, για διεθνείς οργανισμούς, ε, υπηρεσίες κλπ ε, αναφέρονται ως υψηλού κινδύνου. Ε, θα, ε, η στήριξη του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από λιγότερο κίνδυνο. Μπορεί αυτό να δικαιολογείται λόγω των διαφορετικών διαδικασιών, αλλά η δημοσιονομική στήριξη επιτυγχάνει το στόχο της. Εγώ Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ερωτηθούν οι κυβερνήσεις όλων των χωρών που πήραν δημοσιονομική στήριξη ε, να, να κληθούν να δικαιολογήσουν ε, τις δαπάνες αυτές. Ε, πολλές φορές δεν είναι, δεν είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Και εδώ λοιπόν υπάρχει πεδίο για βελτίωση. Τέλος, αν μου επιτρέπει, ακόμα δύο λεπτά να μιλήσω κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Μιλήσατε για την διαχείριση των συνόρων. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μπορεί να έχουμε καλή πρόθεση, αλλά να πετύχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Στο Τσάντ ε, έχω υπόψη πώς έγινε η διαχείριση των συνόρων. Είχαμε δαπανίσει σημαντικά κονδύλια για συνοριακά φυλάκια, για συνοριοφύλακες. 12 ειδικά πλοία κατασκευάστηκαν ε, για τη θάλασσα του Τσάντ ε, και για να ε, λειτουργούν στις ακτές, ως εδώ καλά, αλλά νότιο-δυτικά του Τσάντ οι άνθρωποι είναι κτηνοτρόφοι και πήγαιναν τα ζώα στο, στην Νιγηρία ακολουθώντας ένα δρόμο ο οποίος ήταν πάντα ανοιχτός Τώρα έχει ε, ε, κλείσει γιατί το κράτος του Τσάντ έχει χειροκοπήσει, ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αμείβονται και θέλουν να πάρουν χρήματα για να βοηθήσουν τη διέλευση των ζώων. 160.000 άνθρωποι από την περιοχή του Τσάντ έπρεπε να μετεγκατασταθούν λόγω του Μπόκο τώρα ζουν σε χωριά με άλλους αυτόχθονες και δεν μπορούν να ασκήσουν και αυτή η γεωργική δραστηριότητα μαζί με τους αυτόχθονες, τους ντόπιου. Ε, χρειάζονται λοιπόν να ε, χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Resilience για να αντιμετωπιστούν ε, όλες αυτές οι εντάσεις συγκρούσεις και θα πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες και για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας από όλους και για το, τη σχολική εκπαίδευση θα πρέπει να ε, τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Εμείς είπατε δεν δίνουμε στρατιωτική ε, υποστήριξη. Ε, ε, στο Τσάντ όμως υποστηρίξαμε ένα κτίριο για στρατιωτική εκπαίδευση πολύ σύγχρονο με ηλιακούς συλλέκτες. Είπαν όμως ότι χρειάζονταν και ένα πεδίο βολής ε, και χρειάζονταν και κάποιες, ε, κάποια στήριξη για τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το δώσουμε εμείς, άρα δεν γίνεται και στρατιωτική εκπαίδευση. Ε, έμεινε μισό το έργο. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε από την αρχή για να έχουμε καλύτερους τρόπους συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ε, αναφερθήκατε στο καινούριο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πού πρέπει να συνεργαστούμε. Εμείς ε, υποβάλαμε και γραπτός κάποιες ε, πιο λεπτομερείς ερωτήσεις. Υποβάλαμε γραπτός ερωτήσεις πιο λεπτομερείς και εμείς εδώ στην Επιτροπή θέλουμε η αναπτυξιακή συνεργασία να αποκτήσει τη σημασία που της αρμόζει, να εργάζεται με καλές μεθόδους και να πρικοδοτείται όπως της αξίζει και από τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τσέλερ για αυτά τα συμπερασματικά σχόλια. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο και περνάμε στο σημείο 13. Πρόκειται για το Γενικό Προπολογισμό της ΕΕ για το 8, 1, το 10 και 10 το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Μετά από αυτή την εισβάθος συζήτηση, το προηγούμενο κεφάλαιο θα είμαι σύντομος. Τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Ταμεία χρηματοδοτούν την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής και ε, τα υπερπάντια εδάφη περίπου για 60 χρόνια. Σήμερα η γνωμοδότησή μας για την αξιοπιστία των λογαριασμών και την ε, ε, κανονικότητα των εισόδων για τα ΕΤΑ είναι θετικό, είναι θετική όπως τα προηγούμενα έτη για την νομιμότητα ε, των πληρωμών. Ε, δίνουμε μία αντίθετη νομοδότηση, καθώς οι πληρωμές ε, πλήττονται από λάθη. Το επίπεδο λάθους για τις πληρωμές είναι 3,3% που είναι λίγο μικρότερο από πέρσι. Αν η στήριξη προπολογισμού και η δράσεις ε, των δωρητών αποκλειστούν από το δείγμα, το εκτιμόμενο επίπεδο δράσης είναι 4,4%. Από τις 143 ε, συναλλαγές ε, που ελέγξαμε, 26 είχαν ποσοτικοποιημένα λάθη. Σε δύο περιπτώσεις, από τις 26, η Κομισιόν είχε αρκετές πληροφορίες για να προλάβει να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες αυτές. Σε 10 περιπτώσεις από τις 26 οι συναλλαγές υπόκειταν σε, μια, σε έναν άλλο έλεγχο ή επαλήθευση δαπάνης, όμως ε, και πάλι δεν βρέθηκαν τα λάθη τα οποία βρήκαμε εμείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό λαθών 32% οφείλεται στη μη συμμόρφωση με τους ε, κανόνες για τις δημόσιες συμβάσει. Βρήκαμε περιπτώσεις στι οποίες οι συμβάσει ανατέθηκαν χωρίς ε, να υπάρχει ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής ή δεν ακολουθήθηκαν οι αρχές διαφάνειας και ίση μεταχείρισης ε, στη διαδικασία. Το 2016 η ΓΔ, ο Γενικός Διευθυντής συγγνώμη, της ε, κάλυψε ε, και τις ε, επιδοτήσεις ε, και τις εκτιμήσεις προγραμμάτων υπό την έμεση διαχείριση. Αυτό συνάδει με τις συστάσεις μας και τις παρατηρήσεις μας σε αυτή και σε προηγούμενες αιτήσεις εκθέσεις. Ακόμη και αν ε, το εναπομένον ε, ποσοστό φάλματος ε, εκτιμά ότι το ποσοστό λάθους είναι κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2% πάνω από τις μισές τήσιες δαπάνες υπόκειται σε επιφύλαξη. Ευχαριστώ. Μπορείτε να δώσετε τώρα την απάντησή σας κύριε Πίτροπε και μετά θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εξέτοιμα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, θέλω να ευχαριστήσω την συγκητρία την κυρία Κάπελ που παρουσίασε την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Χαίρομαι που οι περισσότερες από τις συστάσεις ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου από τα προηγούμενα έτη έχουν εφαρμοστεί. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, φετινές ε, συστάσεις η Κομισιόν τις δέχεται και επίσης θα βάλουμε τα δυνατά μας να τις εφαρμόσουμε. Το γεγονός ότι το πιο πιθανό επίπεδο λάθους κατέβηκε από 3,8 σε 3,3% οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο προηγούμενο έργο του ελεκτικού συνεδρίου και στις συστάσεις του που συνεχίζουν να καθοδηγούν τις προσπάθειες των Κομισιόν να βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα ελέγχου. Εγώ ε, δηλώνω εκ νέου την ε, δέσμευσή μου να μειώσω περαιτέρω το ποσοστό λάθους ε, παρά το πολύπλοκο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Όπως υποσχέθηκα, θα ήθελα να επανέλθω στην επιφύλαξη σε σχέση με την διαχείριση του μέσου, του Αφρικανικού μέσου για την ειρήνη. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί όπως ανέφερα η ασφάλεια και η ειρήνη ή η έλλειψή τους έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αναπτυξιακή μας ε, προσπάθεια. Επομένω, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αυτή την επιφύλαξη γιατί παρά σημαντική πρόοδο παραμένουν κάποιοι κίνδυνοι. Συνεργαζόμαστε στενά με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης ε, να ξεπεράσουμε τις ε, αδυναμίες στον έλεγχο που έχουν εντοπιστεί και ε, παίρνουν πολύ σοβαρά τον οδικό χάρτη με τις συστάσεις ε, για να μπορέσουν να περάσουν επιτυχώς μία αξιολόγηση πυλών. Εν τω μεταξύ, μέτρα μετριασμού συνεχίζουν να εφαρμόζονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί στην ε, πιο πρόσφατη αξιολόγηση πυλώνα, ιδίως ε, σε ό,τι αφορά τα λογιστικά συστήματα και τα συστήματα δημοσίων προμηθειών. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την εξάντε έγκριση των ε, σχεδίων ε, για τις δημόσιες συμβάσεις, ε, διαδικασίες μη αντίρρησης για την ανάθεση των συμβάσεων, τις τελευταίες πληρωμές να γίνονται μόνο μετά από θετικά αποτελέσματα ελέγχουν και ενισχυμένους μηχανισμούς παρακολούθησης. Η συνεργασία μας υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να είναι πολύ αποτελεσματική. Και ε, καθώς επικεντρωνόμαστε στην συνεχή παράδοση θετικών αποτελεσμάτων, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την αρχιτεκτονική για καλύτερη ε, διαχείριση επιδόσεων και υποβολή εκθέσεων. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και για τις ε, επικοδομητικές συνεισφορές σας. Ευχαριστώ, κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά το ελεγκτικό συνέδριο και τον Επίτροπο. Σήμερα σημειώνουμε πολλά θετικά. Μείωση του ποσοστού σφάλματος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου ελήφθησαν υπόψη από την Κομισιόν. Ακούσαμε ότι το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3,3, 143 συναλλαγές ελέγχθηκαν, 26 επεκρίθησαν ως ελαττωματικές με σφάλματα και ένα τρίτο του ποσοστού σφάλματος, όπως είπε ο Επίτροπος, έχει να κάνει με την μη τήρηση των κανόνων και γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη παρακολούθηση και πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων και όπως είπε και ο Επίτροπος, ε, για παράδειγμα, εκ θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων έλεγχος των ε, σχεδίων ανάθεσης. Έτσι θα μειωθούν τα σφάλματα που αφορούν στη μη τήρηση των κανόνων ανάθεσης και του χρόνου θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Γενικά ε, θα γίνουν αλλαγές ε, μετά το 2020 και στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι το σημερινό μας θέμα, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου, γιατί θα υπάρξουν αλλαγές. Ε, το Ταμείο είναι το βασικότερο Ταμείο ε, για τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής, ΑΚΕ και των υπερποντίων χωρών και έχει πολλά χρηματοδοτικά μέσα μεγάλης σημασίας για τις χώρες αυτές. Ε, βοήθεια που δεν επιστρέφεται, ε, δανειοδότηση του στον ιδιωτικό τομέα με συμφέροντες όρους. Σημαντικό εδώ και αναφέρθηκε πολλές φορές είναι ότι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των κονδυλίων από το Ταμείο ε, ενισχύει τη συνοχή μεταξύ πολιτικής, αναπτυξιακής πολιτικής και γενικότερων κοινωνικών στόχων, ε, στόχων περιβαλλοντικών, προστασίας κλίματος, ε, ε, μετανάστευσης κλπ. Ο Επίτροπος είπε για τα trust funds και πόσο σημαντικό είναι να ε, πάνε χρήματα και στην διαχείριση των συνόρων που είναι σημαντική παράμετρος για την ενίσχυση της ασφάλειας και το ταμείο, τα, τα καταπιστευματικά αυτά ταμεία ανταποκρίνονται στους σύγχρονους στόχους που έχει μια κοινωνία που ε, αφορούν σε μεγάλο βαθμό σήμερα την μετανάστευση. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη εστίαση εκεί. Στην περσινή έκθεση ο εισηγητής ε, είχε αναφερθεί πολύ και στην καταπολέμηση της φτώχειας σε σχέση με τη μετανάστευση. Αυτό πρέπει να εξακολουθήσει να είναι σημαντική παράμετρος και στην φετινή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επίτροπε, θέλατε να σχολιάσετε. Ε, Ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο, την εισηγήτρια και τον επίτροπο που ήρθε προσωπικά εδώ. Νομίζω ότι ο τρόπος που, με τον οποίο προετοιμάστηκε για την σημερινή συζήτηση δείχνει την σημασία που αποδίδει στα ζητήματα αυτά η Επιτροπή. Μακάρι να ήταν πάντα το ίδιο προετοιμασμένοι όλοι. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ σε κάποια συμπεράσματα του ε, Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Κομισιόν και στις ερωτήσεις μετά στην Κομισιόν. Κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναπούμε χρήση των κονδυλίων από αυτό το ταμείο θα πρέπει να ελέγχονται πάρα πολύ αυστηρά, διότι εδώ ε, υπάρχουν πιθανότητες σφάλματος ή δεν υπάρχει τεκμηρίωση για την καταβολή ε, μισθών. Ε, δεν υπάρχουν πάντοτε τα αποδεικτικά στοιχεία. Ε, το 2016 βλέπουμε να αναδύονται πάλι τα ίδια προβλήματα, όπως κάθε άλλη χρονιά. Κοιτάζοντας την έκθεση τη φετινή και τις προηγούμενες, βλέπω ότι τα ίδια θέματα μπαίνουν ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, στα έσοδα. Το ποσοστό σφάλματος δεν ήταν υψηλό. Έτσι ήταν και στο παρελθόν. Όμως κάποια έγγραφα λείπουν πάντοτε. Έλειπαν ε, παλιά, λείπουν και τώρα. Ε, θα πρέπει να επιμένει ο ελεγκτής, να υποβάλλονται τα σχετικά αποδεικτικά για τη μισθοδοσία. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να ε, προτείνει μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του σφάλματος. Αναφέρθηκε αυτό. Άλλο, συμφωνώ με το ελεγκτικό συνέδριο που λέει ότι η Κομισιόν πρέπει να ελέγχει πιο λεπτομερώς τις ε, δαπάνες. Υπάρχουν ε, ορισμένα έργα που ολοκληρώνονται, ε, οπότε το ποσοστό σφάλματος ε, μειώνεται και γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται πια αυτές. Υπάρχουν προβλήματα με δαπάνες ύψους 303 εκατομμύρι, εκατομμυρίων. Πώς γίνεται αυτό. Θέλετε να απαντήσετε, Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Κάποια από τα ζητήματα που εξετάσαμε για τον προπολογισμό έχουν μια σημασία και σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση των ε, έργων ε, και την εφαρμογή του Ανατοξιακού Ταμείου. Αυτό ισχύει και για την αρρωγή του προπολογισμού, αλλά και των ενεργειών και τη λειτουργία του Κατευθυντικού Ταμείου, γιατί το τμήμα προκύπτει από τα αποτελέσματα EDF. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ ακόμα περισσότερο στις προσπάθειές μας να καλύψουμε αυτή την τελική ευθεία, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την ε, περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος ε, στο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Είναι μεγαλύτερο από ό,τι στον προπολογισμό, Σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης έχουμε καταρτήσει και εγκρίνει ένα ε, σχέδιο δράσης το οποίο θα λαμβάνει υπόψη ακριβώς τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Και με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος για να κατέβουμε από το όριο σημαντικότητα, το οποίο σαφώς είναι και ο στόχος μας. Για κάποιες από τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Αναπτυξιακό Ταμείο, βλέπουμε ότι χάρη στην ευελιξία ορισμένων ε, λειτουργιών και μέσων προβλέπονται από το Αναπτυξιακό Ταμείο, ε, μπορούμε ιδίω στο νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να τα λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, αυτών των ε, προγραμμάτων. Στο EDF έχουμε σημαντικό ποσό, ίσως 20% των 30 δις συνολικά. Περίπου το 20% λοιπόν ε, των ε, αποθεματικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε αναδυόμενες προκλήσεις αλλά και νέες προτεραιότητες. Οπότε δεν έχει μεγάλο νόημα από τώρα ε, να καλύψουμε και να προδικάσουμε πού ακριβώς θα πάνε όλα τα κονδύλια. Θέλουμε λοιπόν αυτή την ευελιξία για το επόμενο ΠΔΠ, ιδίω. και αυτό είναι μια σημαντική δυνατότητα που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω σε ό,τι αφορά την ένταξη του EDF ε, στον προπολογισμό, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι το ένα. Μετά, σε ό,τι αφορά τα πρώιμα ενδεικτικά προγράμματα, τα εθνικά δηλαδή, για, εντός του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου, Είχαμε τώρα, για παράδειγμα, στην Καραϊβική τις τραγικές επιπτώσεις ε, του τυφώνα. Πρέπει λοιπόν πολύ σύντομα και θα είμαστε σε θέση ε, να προβούμε σε ε, ανθρωπιστικές ενέργειες αλλά και πιο μακροπρόθεσμες ε, ενέργειες αύξησης της ανθεκτικότητας από τα αποθεματικά του Ανατοξιακού Ταμείου. Τώρα, με ποια ακριβή διαδικασία θα γίνει αυτό ε, και με την ε, εμπροστοβαρή δηλαδή προσέγγιση και με συμπλήρωση των κονδυλίων στη συνέχεια για να χρηματοδοτήσουμε τις ε, ενέργειες αυτές. Θέλουμε όμως ε, εμείς να διατηρήσουμε αυτή την ευελιξία στα προγράμματα που θα ενταχθούν ε, στο μηχανισμό του επόμενου πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Εμείς έτσι θεωρούμε ότι θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το ταμείο Μια σειρά επιμέρου στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, όταν τελικά αποφασίσουμε την ε, κατάρτιση του προπολογισμού για το Ανατοξιακό Ταμείο. Όμως βλέπουμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εν γέννη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώς ε, και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα είναι σημαντικός εταίρος προκειμένου το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο να διατηρήσει την συνολική του ικανότητα, ισχύ και ευελιξία. Ε, προκειμένου να έχουμε και τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο στους ε, αναπτυξιακούς μας στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Κύριε Ιτάλα, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Εν συντομία, για αυτά που είπε ο κύριος Σετσκόφσκι για τους πολύ αυστηρούς ελέγχους, αλλιώς ε, υπάρχει το ενδεχόμενο απάτη. Συμφωνώ, αλλά πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Τώρα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Χρειαζόμαστε επιτόπιους ελέγχους και το έχω δει από την ε, εκπείρα δηλαδή, ότι δεν φτάνει ε, από το γραφείο μας να κάνουμε τους ελέγχους. Πρέπει να κάνουμε επιτόπιου ελέγχους, όμως βέβαια αυτό πρέπει να, για να γίνει αυτό πρέπει να αυξήσουμε και τη χρηματοδότηση. Σε αυτό συμφωνώ όμως. Ε. Η συγγήτρια, κυρία Κάπελ. Να προσθέσω κάτι. Ε, είναι πολύ σημαντική και σημαντική επιτόπιη έλεγχη. Γιατί ε, το Ταμείο Ανάπτυξης ε, δίνει βοήθεια από τον προϋπολογισμό. Η Κομισιόν σκέφτεται να μειώσει την δημοσιονομική στήριξη μέσα από το ε, Ταμείο Ανάπτυξης διατηρώντας όμως την απαραίτητη ευελιξία για να υπάρχει ευέλικτη αντίδραση το Ταμείο σε ε, προβλήματα όπως τυφώνες κλπ. Μπορεί δηλαδή να μειωθεί η δημοσιονομική στήριξη και να παραμείνει το Ταμείο ευέλικτο. Θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ αυτή την ερώτηση. Ναι, η ευελιξία του ΕΤΑ είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του μέσου και σίγουρα θέλουμε να το διατηρήσουμε. Όμως αυτό είναι ένα κοινό εγχείρημα. Είναι κοινή αποστολή μας, ε, θα έλεγα, να διατηρήσουμε την ευελιξία στους ε, χρηματοοικονομικούς κανονισμούς ε, που καταρτίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά θέλουμε και να διατηρήσουμε τη συνολική ικανότητα να έχουμε ένα κατεπιστημιακό ταμείο και συναλλαγές που θα υπόκειται σε καλό έλεγχο και σε διαφάνεια. Ένα σημαντικό τμήμα της εφαρμογής του ΕΤΑ είναι μέσω project που στηρίζεται από τον προπολογισμό. Τώρα, η στήριξη είναι 20-30% του συνολικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Θα ήθελα να διατηρήσω το επίπεδο αυτό, αλλά να βελτιώσω την ικανότητά μας των κριτηρίων εξπόστη και εξάντως προς την παρακολούθηση και της διατήρησης ε, του διαλόγου πολιτικής με τις χώρες εταίρους ως προς την εφαρμογή όλων των κριτηρίων ε, ή των προηγούμενων κριτηρίων που χρειάζεται για να δοθεί ο επόμενος ε, γύρος ε, δημοσιονομικής στήριξης. Θέλω τώρα λοιπόν να ενδυναμώσω τη συνεργασία μας για να θεσπιστεί το ορθό κανονιστικό πλαίσιο, ο σωστός χρηματοδοτικός κανονισμός που θα καταστήσει ε, τις ε, δράσεις ε, του ΕΤΑ αλλά και τις δράσεις δημοσιονομικής στήριξης πιο κατάλληλες και πιο κοντά στο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Επίτροπε. Είχα μια συνάντηση με 100 Γάλλους επιχειρηματίες και έπρεπε να βοηθήσω. Ε, και ο, ε, ο, κύριος Τσέλερ. Ευχαριστούμε. Το ΕΤΑ είναι περιορισμένο και χρονικά, αλλά και η περιφερειακή του αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένη. Είναι ένα θεμέλιο ε, για τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ. Ε, ακολουθεί τη Συμφωνία Κοτονού, αλλά το 2020 αυτή τελειώνει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Συμφωνία του Κοτονού και αν θα υπάρχει το ΕΤΑ όπως είναι τώρα. Είναι ένα ειδικό ταμείο, δεν είναι κομμάτι του προϋπολογισμού. Τι βλέπει η Κομισιόν να γίνεται στο μέλλον με τη Συμφωνία Κοτονού Αφενός και τι δυνατότητες και τι κονδύλια θα έχει το ΕΤΑ. Υπάρχει η προοπτική αν δεν συνεχιστεί η Συμφωνία Κοτονού αυτά τα κονδύλια να περιοριστούν και να πάνε για αναπτυξιακή πολιτική μέσα από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να μην εφαρμόζεται μόνο για τα 72 ε, κράτη ΑΚΕ, αλλά να αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική γενικότερα. Πρέπει να συζητήσουμε πολύ το θέμα αυτό βέβαια για να πιστούν όλα τα κράτη-μέλη, αλλά σίγουρα η συζήτηση αυτή είναι απαραίτητη. Yes, Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση. Συμφωνώ πλήρως. Αυτή τη στιγμή δεν ε, έχουμε μια ξεκαθαρή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί το πλαίσιο της συνεργασίας μας μετά το κοτονού. Ούτε έχουμε σαφή εικόνα για, πώς ε, θα μοιάζει, για το πώς θα μοιάζει το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης μετά το 2020, αφού λήξει το ποδίπου. Τουλάχιστον για μένα όμως ε, υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία όταν μιλάμε για τις διευθετήσεις μετά το κοτονού. Μαζί με τα κράτη-μέλη αλλά και σε συνεργασία με τους εταίρους μας στις χώρες ΑΚΕ, ερχόμαστε πιο κοντά στο να διαμορφώσουμε την ε, νέα εταιρική σχέση, την συμφωνία εταιρική σχέσης μετά το Κοτονού, η οποία θα είναι πιο συγκεκριμένη ως προς τις περιφέρειες αλλά θα κρατήσει και όλα τα θετικά στοιχεία της σημερινής συμφωνίας, δηλαδή το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που θέλουμε να προωθήσουμε με τις χώρες εταίρους. Η ιδέα λοιπόν είναι από την πλευρά της Κομισιόν να παρουσιάσουμε το Δεκέμβρη ε, μία, ένα σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για τη συμφωνία που θα ακολουθήσει, που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού ουσιαστικά θα μιλάμε για μια συμφωνία καθολική που θα κρατά αυτές τις βασικές αξίες στη συμφωνία μας και κατόπιν θα έχουμε τρεις περιφερειακούς πυλώνες για την Αφρική, για τις χώρες της Καραϊβικής αλλά και για τον Ειρηνικό και εκεί θα ε, καθορίζουμε πώς θα δημορφωθούν οι εταιρικές μας σχέσεις στον πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό τομέα με τις χώρες αυτές. Όμως σκοπεύουμε να κάνουμε μια αποσύνδεση, δηλαδή να διατηρήσουμε τις διαπραγματεύσεις για το νομικό πλαίσιο ξεχωριστά από τα χρηματοδοτικά κονδύλια που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε στην πράξη τη μελλοντική συμφωνία με το τοκοτουνό. Αυτό το κάνουμε γιατί το θέμα της ένταξης στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ είναι μια επιλογή είναι ίσως η πιο σοβαρή επιλογή για το μέλλον. Όμως θα πρέπει να συζητήσουμε και με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη το πώς η συμπερίληψη του Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό θα αντιμετωπίσει το ανώτατο όριο που έχει συμφωνηθεί του 1% για τις πληρωμές, του 1,2% του ΑΕΠ ε, για τις επιστώσεις ανάληψης ε, υποχρεώσεων. Δηλαδή, το, πρέπει να σκεφτούμε και τα νότατα όρια του προϋπολογισμού, πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα του Brexit ε, και τι θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα καταβάλει κονδύλια ή όχι στον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι σημαντικό. Και υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να δούμε. για το πώς θα έχουμε αναπτυξιακά μέσα με το ΕΤΑ εντός προϋπολογισμού που θα συνεισφέρουν στην συλλογική δέσμευση που έχουμε αναλάβει στο να φτάσουμε το στο 0,7 του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί η συμφωνία με το Κοτονού, αλλά και πώς θα διαμορφωθεί και η δική μας χρηματοδοτική ικανότητα με τη συμπερίληψη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Α, η κυρία Γιάλα Ζέντερ. Λυπάμαι Ήμουν ε, στην Επιτροπή Μεταφορών και καθυστερήσαμε πολύ με τις ψηφοφορίες. Λυπάμαι κύριε Επίτροπε που δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Είχα δύο μικρές ερωτήσεις. Έχουν να κάνουν με το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. δηλαδή στο τμήμα που παρεμβαίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης με σημαντικά κονδύλια. Θέλουμε να ξέρουμε το εξή. Πώ μπορούμε να ελέγξουμε ήδη εντό του καταπιστευματικού ταμείου συγκεκριμένε δραστηριότητε που σχετίζονται, παραδείγματο χάρη, με τον έλεγχο των συνόρων και συνεπιφέρουν στο καταπιστευματικό ταμείο αστυνομικέ δραστηριότητε, και πιο κατασταλτικού τύπου, να το πω έτσι, ε, πέρα δηλαδή από τις ε, καθαρές δράσεις ανάπτυξης ε, και συνεργασίας. Ε, δηλαδή, ναι, εφόσον το ΕΤΑ συμμετέχει στο Καταπιστηματικό Ταμείο, πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε ότι οι δραστηριότητες ε, αυτές που εντάσσονται στο καταπιστευματικό ταμείο δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του ΕΤΑ. Και κάτι ακόμα σε σχέση με τις ε, συνεισφορές στο καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. Βλέπουμε ε, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα κριτήρια, δηλαδή αν ένα κράτος μέλος μπορεί να παρέμβει με έναν απεριόριστο τρόπο Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσουμε και γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ρωτούσαμε γιατί έχει περισσότερο ε, ενδιαφέρον ή συμφέρον να το κάνει μια χώρα αυτό. Δηλαδή, πόσοι ε, τώρα αξιολογεί τα ποσοστά συμμετοχή στο κρατών μελών, μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή. Γιατί είναι ιδιαίτερα άνηση η συμμετοχή αυτή Μπορεί κάποια μια άνηση συμμετοχή, δηλαδή και αν αυτή που μπορεί να είναι πολύ ψηλή, να επιφέρει ένα είδου ελέγχου, εντολή. Δηλαδή έχουμε διάφορες ε, χώρες ε, που μπορεί να έχουμε άνηση συμμετοχή, αυτές που συμμετέχουν περισσότερο. Ποια είναι τα κριτήρια που διέπουν αυτή τη συμμετοχή. Δηλαδή πρέπει να δούμε αν ένας κράτος μέλος ε, ε, μπορεί να συνεισφέρει χωρίς κάποιο όριο. Θα έλεγα πως όχι, γιατί αυτό ε, ουσιαστικά μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις. Θα ήθελα να μου πείτε πώς η Κομισιόν το έχει θεσπίσει αυτό. Yes, thank you very much for this. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας, για τις λειτουργίες ε, του Καταπιστευματικού Ταμείου το συζητήσαμε προηγουμένως όταν εξετάσαμε τον προλογισμό, αλλά αντίστοιχα σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση και τον έλεγχο των συνόρων που χρηματοδοτείται από ε, αυτές τις λειτουργίες. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι το Καταπιστευματικό Ταμείο ουσιαστικά δεν χρηματοδοτεί τον έλεγχο των συνόρων με τη στενή έννοια του όρου, αλλά περισσότερο αφορά τη διαχείριση συνόρων. Λειτουργίες δηλαδή που θέλουμε να ενισχύσουμε σε ορισμένες από τις χώρες εταίρους μας. Όμως πάντα θέλουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητές τους ε, για τη διαχείριση συνόρων, αλλά με ήπια μέσα. Δεν θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε το, τις θεωρητικές τους δυνάμεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε πάντα να δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες από τις καταπιστευματικές μας ενέργειες, θα πρέπει να μπορούμε να την παρουσιάσουμε ως επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον έλεγχο των συνόρων, καλό είναι οι χώρες εταίροι να απευθύνονται στα κράτη-μέλη και όχι σε εμά μέσω του καταπιστευματικού ταμείου. Φυσικά και με βάση τη συνθήκη δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε στρατηγική ικανότητα κτλ. Αλλά θέλουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο είτε από το Καταπιστευματικό Ταμείο είτε από τις ε, ενέργειές μας μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης. Για τη συμμετοχή των κρατών μελών στα καταπιστευματικά ταμεία. Στην αρχή η προσέγγιση μας ήταν λίγο πιο γενική. Πιέζαμε ακόμη περισσότερο τα κράτη-μέλη να ισοσκελίσουν τη δική μας ε, συνεισφορά στα καταπιστεύματα, ιδίως αυτό της Αφρικής. Όμως αυτή η γενική έκκληση προς ε, συμμετοχή δεν είχε και την ανάλογη ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη. Στο ποσοστό δηλαδή των ε, συνεισφορών ε, ε, της δικής μας ενισφοράς ε, στα ταμεία αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των κρατών μελών. Τους καλέσαμε, τα καλέσαμε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε ίσο επίπεδο με εμά και μας απάντησαν κάποιες φορές ότι έτσι κι αλλιώς συμμετέχουν γιατί τα δικά τους χρήματα είναι που πηγαίνουν και στον περιπολογισμό και στο Ταμείο Ανάπτυξης. Επομένως, Τώρα έχουμε κάπως προσαρμόσει την προσέγγιση μας. Θα θέλαμε να πούμε ότι την έχουμε βελτιώσει. Θέλουμε πραγματικά ε, να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη πώς μπορούν να συμβάλλουν, όχι μόνο σε ό,τι αφορά με την γενική του συνεισφορά στο, ε, στις πληρωμές, στα καταπιστευματικά ταμεία, αλλά πώς θα συμβάλλουν σε πιο συγκεκριμένα ε, μεμονωμένα προγράμματα που έχουμε αναπτύξει. Για παράδειγμα, έχουμε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα στη Λιβύη και στον Ήγυρα, όπου ε, βοηθούμε ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την οικειοθελή επιστροφή των ε, μεταναστών και την επανεισδοχή τους, μάλλον την επανένταξή τους στην χώρα προέλευσής τους. Αυτό το πρόγραμμα με αυτούς τους συγκεκριμένους δηλαδή εταίρους πιστεύουμε και μάλλον βλέπουμε ότι είναι πιο σκόπιμο να συμμετάσχουν εκεί τα κράτη-μέλη και είναι και πιο πρόθυμα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν εκεί. Άρα Αυτή δηλαδή η συνεισφορά σε συγκεκριμένα προγράμματα θα ενισχύσει και τη συνολική συμβολή των κρατών μέλων. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια σύντομα. ...3,3 ποσοστό σφάλματος. Πρέπει να μειωθεί κι άλλο κυρίως μέσα από καλύτερη παρακολούθηση των κανόνων ανάθεσης και έγιναν σχετικές προτάσεις. Αυτός είναι ο στόχος, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ευελιξία. Και οι δύο μεγάλες προκλήσεις στο ΕΤΑ είναι η αλλαγή από το 2020 στο δημοσιονομικό πλαίσιο και η συνέχεια του Κοτονού δύο μεγάλες προκλήσεις και παράλληλα ο στόχος της περαιτέρω μείωσης του ποσοστού σφάλματος. Ακόμα χρειάζεται πολλή δουλειά. Ωραία. Ε, αυτό το είχε πει και ο Επίτροπος. Προχωρούμε. Ε, ο κύριος Λαζαρόλη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να έρθουμε και να σας δώσουμε μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της τράπεζας στις χώρες ΑΚΕ. Εστιάζουμε στο τι επέτυχε πέρσι, το 2016 η τράπεζα. Οι βασικές προτεραιότητες στην περιοχή βέβαια παραμένουν οι ίδιες. Επιτρέψτε μου να τονίσω τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων και τους βασικούς στόχους της τράπεζας και που είναι η ανάπτυξη του ε, δημοσίου τομέα, η ανάπτυξη βιώσιμης ε, υποδομής, δράση για το κλίμα, αύξηση 35% των δανείων μέχρι το 2020, περιφερειακή ολοκλήρωση. Αυτά είναι όσα προσπαθούμε να κάνουμε ως τράπεζα. Ο γενικός στόχος είναι βέβαια η μείωση της φτώχειας. Καθαρά ποσοτικά η δραστηριότητα πέρσι ήταν σχετικά σταθερή, αν συγκριθεί με το 2015 είχαμε μικρή πτώση ε, από, 930, από 936 πήγαμε στα 915 ε, αλλά αυτό η μείωση των πιστώσεων αντισταθμίστηκε στην αύξηση των εγκρίσεων που είναι από 1,05 δις το 2015 στο 1,3 δις το 2016 και σημειωτέων ε, είχαμε πολλές ε, εκταμιεύσεις που έφτασαν σε 947 εκατομμύρια έναντι 538 ευρώ. Γενικά, αν δούμε το χαρτοφυλάκιο των ε, πράξεων, των επιχειρήσεων, θα δείτε ότι το μέγεθος των μεμονωμένων έργων μειώνεται και γι' αυτό, παρά τις μειωμένες πιστώσεις, τα έργα έμειναν στο σταθερό αριθμό των 29 και επιμερίζονται μεταξύ ΕΤΕ ή το φάκελο των ιδίων πόρων. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η αύξηση ε, μιας υποσυνιστώσας του χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις. 11 έργα υποστηρίχθηκαν από εκεί, από και 97 εκατομμύρια, που είναι ένα ποσό ρεκόρ. Θα θυμάστε ότι αυτός ο φάκελος δημιουργήθηκε το 2015, ο ε, ε, φάκελος χρηματοδότησης αντικτύπου χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη του, της δέσμης μετανάστευσης ΑΚΕ που δημιουργήθηκε το 2016 στην τράπεζα που είναι το καλύτερο παράδειγμα της προσαρμοστικότητας και της ε, ευελιξίας της ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτή η δέσμη πάει να καταπιαστεί με τη ρίζα του κακού της μετανάστευσης στην υποσαχάρια Αφρική. Ε, εφιστώ την προσοχή σας ε, στο μέγεθος της προσπάθειας. 200 εκατομμύρια πρόσθετη πόρη ε, στα πλαίσια του Impact Financing Envelope. Αυτά είναι κονδύλια που δεν έρχονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό ή τα κράτη-μέλη. Ε, αυτά είναι ανακυκλούμενα κονδύλια που επαναχρησιμοποιούνται για νέα project και νέα έργα. Και άλλα, ε, ε, εκτός από αυτά, 500 εκατομμύρια από το επενδυτικό μέσο πάει σε έργα για το δημόσιο για να καταπολεμηθεί η μετανάστευση. από δύο στα 2,5 δις πήγαμε τα... η δέσμη αυτή ε, υλοποιείται ήδη. Θέλουμε να αναπτύξουμε ε, ευκαιρίες ε, επικεντρωνόμενοι στις, στους νέους και στις γυναίκες, στις δημόσιες υπηρεσίες και έχουμε στόχο χώρες που είναι χώρες διέλευσης και τελικού προορισμού και χώρες προέλευσης. Είναι πολλά τα ε, έργα θα αναφέρω ε, ορισμένα από αυτά που υπάρχουν σε αυτή τη δέσμη για να σας δώσω μια γεύση του τι κάνουμε. Τρία θα αναφέρω. Το ένα είναι η ε, επέκταση στο Καμερούν του συστήματος ηλεκτροδότησης, όπως και στο Κονγκό. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα συνδέσει 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους που στη χώρα στις χώρες αυτές που χρησιμοποιούν ε, λύσεις διαφορετικές, κυρίως βασισμένες στην ηλιακή ενέργεια. Ε, 300 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ήπειρο αυτή δεν έχουν σύνδεση με την κινητή τηλεφωνία. Αυτό είναι για την κινητή τηλεφωνία. Ε, υπάρχει και η πρωτοβουλία για την Αφρική που είναι μια κοινή πρωτοβουλία μαζί με την Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων δηλαδή ADB και η EIB, η δική μας τράπεζα επενδύσεων, 300 ε, εκατομμύρια διατίθενται. Ε, αυτό είναι ένα υπερταμείο το οποίο, ένα fund of το οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις το οικοσύστημα το υποσαχάριο. Και πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες γίνονται για την οικοδόμηση ικανοτήτων. Ένα άλλο project είναι στη Σενεγάλη, ε, αφορά την παραγωγή ρυζιού και την αποθεματοποίηση ε, σε μια χώρα που εισάγει 80% των, του, των αναγκών της ερίζη. Στην Καραϊβική ε, επίσης έχουμε έργα. Θα ήθελα να σας πω τι έκανε η τράπεζα εκεί το 2016. Έχουμε ένα ειδικό μέσο αντικτύπου που δημιουργήθηκε το 2015 Πέρσι ε, δώσαμε πιστώσεις στη Τζαμάικα και τη Δομινικανή Δημοκρατία για μικροπιστώσεις. Αυτό είναι ένα μέσο που πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει πάνω από 100.000 ανθρώπους, ε, χορηγώντας ε, μικρά δάνεια, πολύ μικρά καμιά φορά, χωρίς εγγύηση, και έτσι χρηματοδοτούνται άνθρωποι που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ε, στη Γαλλική Πολυνησία δώσαμε 8,4 εκατομμύρια, κυρίως για επιχειρηματίες και τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες στο νησί. Τώρα, γενικότερα ε, νούμερα, ε, για να σας δείξω γενικότερα τι κάνει η τράπεζα. Οι συνολικές πιστώσεις από τις συνολικές 254 πήγαν στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από αυτές, 210 εκατομμύρια ε, υποστήριξε ΜΜΕ και 44 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για μικροπιστώσεις. 56 εκατομμύρια δαπανίσαμε σε 5 χωριστά equity funds θεωρώντας ότι θα δημιουργηθούν έτσι 2.000 θέσεις εργασίας στις διάφορες εταιρείες όπου κάναμε επένδυση. Ε, από τους ιδίους πόρους μας, που είναι ο δεύτερος πυλώνας που μας επιτρέπει να ε, παρεμβαίνουμε, στηρίξαμε αρκετά τέτοια έργα ε, για την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες που αφορούν την ποιότητα ζωής, 100 εκατομμύρια δολάρια για την ηλεκτροδότηση και πάλι είχαμε κάποια σημαντικά έργα που στηρίξαμε στη Μαδαγασκάρη και σε Νεγάλη ε, για νερό ε, και υγειονομικά μέτρα στον υγειονομικό τομέα και ε, αντιμετώπιση των πλημμυρών. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις πέρα από τα επιμέρους έργα που στηρίζουμε. Να υπογραμμίσω ότι η τράπεζα συνεχώς προσπαθεί να αυξήσει τον αντίκτυπο των εργασιών της, των πράξεών της. Το κάνουμε αυτό παρακολουθώντας τα αποτελέσματα, ε, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το κάναμε και πέρσι ε, με μια νέα εταιρική σχέση με το Παγκόσμιο Αναπτυξιακό Δίκτυο που μας επιτρέπει καλύτερα να παρακολουθούμε τον αντίκτυπο των επιχειρήσεών μας, των δράσεών μας. Ε, χρησιμοποιούμε ερευνητέ και από τις χώρες ΑΚΕ. Θα μπορέσουμε έτσι να αντλήσουμε διδάγματα, να βελτιώσουμε τη δική μας αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα. Δεύτερη παρατήρηση. Βεβαίως και θέλουμε να ε, αυξήσουμε την συμπληρωματικότητά μας, την ευθυγράμμισή μας ε, με τις ε, ενωσιακές πολιτικές, παγκόσμια στρατηγική κλπ. Αυτό ισχύει και για την περιοχή ΑΚΕ, όπου αναπτύσσεται το σχέδιο εξωτερικής αναπτυξιακής δράσης, που θα συζητηθεί για το χώρο της Αφρικής το Δεκέμβρη. Τέλος, συζητήσαμε και προηγουμένως αναφερθήκατε και στο Κοτονού, με την περίοδο μετά το Κοτονού κλπ. Η τράπεζα θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο στη νέα εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ πέραν του 2020 και θέλει να συμμετέχει στις συζητήσεις που θα γίνουν για τη μελλοντική αρχιτεκτονική των σχέσεων αυτών θεωρούμε ότι είναι ε, καταλητικό το μέσον της ε, ε, χρηματοδότησης επενδύσεων. Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε τον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή. Είμαστε πεπισμένοι ότι το ευρωπαϊκό μέσον επενδύσεων είναι ε, πάρα πολύ σύγχρονο, αποτελεσματικό, με ανακυκλούμενα κεφάλαια. Δεν χρειάζεται να δώσουμε καινούριε χρηματοδοτικές ε, εισφορές γιατί ανακυκλώνει τα κεφάλαια ε, για να χρηματοδοτήσει τις γραμμές του προϋπολογισμού του και αν δούμε την μόχλευση αυτών των πόρων βλέπουμε ότι από το 2003 για ένα ευρώ συμβολήσα από το ΕΤΑ είχαμε στηρίξει περίπου 9 ευρώ επενδύσεων. Και αυτή η μόχλευση θα αναμένεται να αυξηθεί μέσα από την επαναχρησιμοποίηση. Μέχρι το 2015 η μόχλευση από τα 9 θα πάει στα 15 ευρώ. Η ευελιξία του χρηματοδοτικού μέσου μας επιτρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τις δραστηριότητές μας στην περιοχή. Δεν περιοριζόμαστε σε αιτήσια βάση, αλλά χαράζουμε μακροπρόθεσμες πολιτικές ε, ε, παράλληλα με τις ε, προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σταματώ εδώ για να προλάβουμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, από το 1 στο 9 η αύξησή μας, η μόχλευσή μας δείχνει πόσο σημαντική εκό είναι το καθήκον και η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, σε σχέση με το Ταμείο. Η Τράπεζα ε, δίνει 2,5 δις, δηλαδή 8% του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου. Και αν αυτό το 8% ε, χρησιμοποιηθεί με χαμηλό ή δυνατόν ε, ποσοστό σφαλμάτων. Ε, αυτά είναι μέσα από τράπεζα. Θα μειώνεται λοιπόν το ποσοστό σφάλματος, έτσι αναμένεται. Από το 3,3 αν μειωθεί θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, με λιγότερα σφάλματα. Και η Τράπεζα Επενδύσεων έχει ιδιαίτερη αξία εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική η συνεργασία με τις Αφρικανικές Αναπτυξιακές Τράπεζες. Αναφέρθηκε συγκεκριμένο project, το Boost Africa Initiative, ε, μαζί με την Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός μοχλός ούτω ώστε να δαπανώνται στοχευμένα και αποτελεσματικά τα κονδύλια του ΕΤΑ. Η μείωση της φτώχειας είναι ο υπέρτατος στόχος, όλα τα άλλα είναι από κάτω. Οι τρεις, ε, ε, η βελτίωση του ιδιωτικού τομέα, βελτίωση υποδομών, ε, προστασία του κλίματος, 25% αύξηση των δανείων, αυτοί οι υποστόχοι έχουν άμεση σχέση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι στόχοι βοηθούν και τις λύπτριες χώρες να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Δώσατε συγκεκριμένα παραδείγματα, πολύ σημαντικά. Επέκταση των τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων, βελτίωση βελτίωση ε, των τηλεπικοινωνιών στο Καμερούν, στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Τζαμάικα, οι μικροπιστώσεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά μέτρα ε, που έχουν ε, σχέση με την μετανάστευση και είναι σημαντικά όχι μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά την καταπολέμηση των αιτίων της μετανάστευσης. Και επίσης, είπατε κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ, την συμφωνία ε, του 2016 για τη μετανάστευση με τις χώρες ε, ΑΚΕ. Και το Impact Financing Envelope ε, παίζει μεγάλο ρόλο. Ελπίζω τα 300 εκατομμύρια να αυξηθούν. Είναι πολύ σημαντικό το μέσον αυτό για να μετριάσει τις μεταναστευτικές πιέσεις και να μειώσει και τα αίτια της μετανάστευσης. Και αν η μόχλευση είναι τόσο υψηλή, τότε χρησιμοποιούνται πολύ καλά τα κονδύλια και ενδεχομένως στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο θα μπορούσαμε να αυξήσουμε και εμείς ε, τα κονδύλια που διαθέτουμε ούτω ώστε να υλοποιούνται από τις τράπεζες ε, αξιόλογα έργα. Ο κύριος Τσέλερ, ευχαριστώ για την ετήσια έκθεση που περιέχει ενδιαφέροντα έργα, χρήσιμα έργα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την τράπεζά σας. Ε, είπατε ότι 30 εκατομμύρια δώσατε στην ε, Εθνική Τράπεζα του Μαλάουι για να αυξήσει την ε, δυνατότητα αποθεματοποίησης γεωργικών προϊόντων. Χρήσιμο πολύ αυτό βέβαια, ιδιαίτερα ε, λόγω της διαφοράς στις εσοδίες κάθε φορά. Η ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Μαλάου είναι από τις πιο διεφθαρμένες Πώς μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα 30 εκατομμύρια θα πάνε σε αυτή τη χρήσιμη επένδυση και δεν θα ε, μπουν στις τσέπες διαφόρων. Ε, σε άλλες χώρες της Αφρικής αυτές δημιουργούνται αποθηκευτικές ικανότητες αλλά τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται δεν ταιριάζουν με αυτά που χρειάζονται για την Αφρική. Και εγώ θέλω να πω κάτι για, το, για τη μόχλευση, για το leverage ένα προς 9. Πόσο κομμάτι είναι ιδιωτικό κεφάλαιο από αυτή τη μόχλευση. Αυτά τα 9 δηλαδή ευρώ από πού προέρχονται, από ποια ιδρύματα. Είναι ε, δημόσιο χρήμα ή και ιδιωτικό. Υπάρχουν ιδιωτικές τράπεζες που συμμετείχαν ή συμμετέχουν. Δεύτερον, πώς επιλέγετε τα έργα ε, μας παρουσιάσατε διάφορα έργα και σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος κατάλογος έργων, πόσο μακροσκελής είναι. Υπάρχει κατάλογος έργων που είναι σε αναμονή. Και η κυρία, Α, η κυρία Γιάλα Ζέντερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων για την παρουσίασή του από το ιστορικό της συζήτηση ε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και για τα σχέδια ανάπτυξης, ένα από τα πολύπλοκά θέματα που είχαμε σκεφτεί όταν θέλαμε να ιδρύσουμε και μία μεσογειακή τράπεζα στην Τινησία. Ε, ήταν όλο αυτό ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει και στα Εθνικά Κοινοβούλια, στη συζήτηση με την ΕΤΕΠ, το πρόβλημα πάντοτε ήταν ότι η τράπεζα είναι ένα μέσο που είναι εκπληκτικό και λειτουργούσε πάρα πολύ καλά για τα μεγάλα έργα, για τις μεγάλες υποδομές ή για τις μεγάλες υπηρεσίες. Όμως ε, σε επίπεδο ε, μικροχρηματοδότησης όπου χρειάζεται να δώσουμε χρηματοδότηση σε ομάδες, το χάρη με προβλήματα όπως οι γυναίκες που υποστηρίζουν τις οικογένειες και ουσιαστικά πρέπει να τις βοηθήσουμε ε, να πουλήσουν κάτι που έχουν καλλιεργήσει στον κήπο τους, ε, παραδείγματος χάρη. Υπήρχε λοιπόν πάρα πολλέ δυσκολίε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το θέμα τη μικροχρηματοδότηση. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έκανε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να σχεδιάσει συγκεκριμένα προγράμματα για τη μικροχρηματοδότηση. Όταν βλέπω τον κατάλογο που μας δώσατε και σας ευχαριστώ πολύ γιατί βλέπουμε εδώ και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί αλλά και τον κατάλογο των ε, πιστοντικών ε, γραμμών ε, των τελευταίων χρόνων, παρατηρώ με κάποια ανησυχία ότι ακόμη και αν έχουν υπογραφεί πολλές συμβάσεις και μιλάω για το ιστορικό 2003-2016, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν δοθεί με τα χρήματα και έχουν ε, γίνει εφαρμογέ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλέ στήλε που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση σε διάφορε χώρε όπου βλέπουμε μηδενικό ποσό. Και παρόλο που έχει υπογραφεί η, σύμβαση, η σύμβαση, δεν υπάρχει κανένα ίχνος εφαρμογή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Τράπεζα Επενδύσεων. Για το θέμα αυτό βλέπω τη λείπει η γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό και πώς σκοπεύετε να το λύσετε. Γιατί εδώ στη χαρακτηματοδότηση πετυχαίνουμε οι οικογένειες, αλλά και άλλες ομάδες, ναι, οι νέοι παραδείγματος χάρη, να μπορούν ε, να επιβιώσουν και να εφαρμόσουν αυτή την ε, μικροοικονομία που αποτελεί τη βάση των κοινωνιών στην Αφρική. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν και πώς ε, θα λύσετε αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε εδώ και εμφανίζονται και στις ε, στήλε. Ο κύριος Λαζαρόλη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα αντιδράσω σε κάποια από τα σχόλιά σας. Να ξεκινήσω με την ε, αλλαγή της ε, φύσης ε, του επενδυτικού ταμείου. Είναι ένα ουσιαστικό σημείο. Έχει να κάνει με το επίκεντρο της λειτουργίας του μέσου. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πρικοδότηση και ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα ποσό που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε έργα περίπου έχουμε 800 εκατομμύρια το χρόνο, ακόμη και μετά το 2020, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουμε ε, στο να ζητήσουμε νέα κονδύλια από τα κράτη-μέλη ή από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτό είναι σημαντικό. Για τον γεωργικό τομέα. Αυτός είναι φυσικά ένα μέσο που η τράπεζα έχει προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Αν δείτε την πραγματικότητα σε κάποιες χώρες, παραδείγματο χάρη στην ε, Σενεγάλη, θα δείτε ότι υπάρχει εισαγωγή ρυζιού κατά 80%. Βλέπετε λοιπόν πόσα πολλά πρέπει να γίνουν ε, σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα με τις μικρές και μισές επιχειρήσεις, τη χρηματοδότηση κτλ. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα κάνει περισσότερα η τράπεζα και στο μετανάστευση ε, θα δείτε ότι εργαζόμαστε τώρα σε περισσότερα πακέτα για τα οποία θα σας υποβάλουμε και εκθέσεις. Τώρα, τα ιδιωτικά κεφάλαια ε, το κάνει αυτό η τράπεζα σε σχέση και με τον αντίκτυπο που έχει ο χρηματοδοτικός ε, κεφάλαιος. Αναφέρθηκα στα 56 εκατομμύρια επενδύσεων ε, νέων πιστώσεων σε αυτά τα πέντε ταμεία. πρόκειται ουσιαστικά για χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από αυτό το συγκεκριμένο μέσο. Αυτά τα ταμεία συνήθως δεν καλύπτουν όσα χρειαζόμαστε για τις επενδυτικές εταιρείες και ε, το ίδιο όπως δεν δίνεται το 100% των πόρων ε, των ταμείων. Έτσι λοιπόν, εμείς ε, παίζουμε ένα ρόλο επενδυτή, anchor investor, Δηλαδή, ήδη πρέπει να υπάρχει κάποιος επενδυτής με καλή φήμη. κοιτάζουμε αν γίνονται σεβαστές οι αρχές στη δραστηριότητα των ταμείων αλλά πέρα από αυτό που συνεισφέρουμε εμείς, πέρα από εμά, θα υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Και αυτή είναι η όλη ιδέα. Η ιδέα είναι να αναπτύξουμε τον χρηματοοικονομικό τομέα στις περιοχές αυτές. Το ίδιο τώρα το Ταμείο ίδιο Κεφαλαίων, όταν χρηματοδοτεί διάφορα έργα, θα το κάνει μαζί και με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν, η ιδέα εδώ είναι να γεφυρώσουμε αυτό που θεωρείται κενό και στη συγκεκριμένη περίπτωση του χρηματοοικονομικού τομέα να αναπτύξουμε μία πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Θα θέλαμε να δούμε ανάπτυξη τα επόμενα έτη μιας τυπολογίας ε, επαγγελματιών όπως ε, παραδείγματος χάρη διαχειριστές ε, ταμείων, κονδυλίων ή νομικών που θα μπορούσαν ε, να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση αυτών των ταμείων. Πώς επιλέγουμε τα διάφορα προγράμματα. Έχουμε διαδικασίες και σε ό,τι αφορά την επιλογή των προθητών αλλά και των ίδιων των σχεδίων. Κάνουμε ε, κάποιους ελέγχους ε, ακαιρεότητας ε, για τους προθητές και κάποιους ελέγχους για τους πελάτες, αλλά φυσικά βλέπουμε και τα ίδια τα προγράμματα, τα ίδια τα έργα, και αυτό όχι μόνο από εντελώς οικονομική σκοπιά, δηλαδή αν ένας προθητής μπορεί τελικά ε, να επιστρέψει τα κονδύλια, αλλά βλέπουμε και την οικονομική πτυχή του project. Είναι ε, ουσιαστικά καλό το project και θα έχει τα απαραίτητα αποτέλεσμα για να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό ε, έχει να κάνει με την αξιολόγηση του σχεδίου. Δηλαδή βλέπουμε τον αντίκτυπο αυτών των σχεδίων και πριν κάποια χρόνια, βάσει και σχολείων που λάβαμε από τους διάφορους διαχειριστικούς φορείς, ένα ε, πλαίσιο μέτρησης το οποίο ακριβώς να μπορεί εκ των προτέρων να καθορίσει ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και στη συνέχεια να τα συγκρίνουμε με αυτό που βλέπουμε ότι γίνεται επί έτσι λοιπόν, ε, αυτό είναι πάντοτε κάτι θετικό γιατί είτε μας βοηθά ε, να μάθουμε, να αντιλήσουμε διδάγματα ή μας βοηθά να έχουμε ένα διάλογο με τους σχεδιαστές του προγράμματος. Η μικροχρηματοδότηση είναι ουσιαστικά κάτι πολύ σημαντικό είναι κάτι που τυπικά υποστηρίζουμε ε, σε ό,τι αφορά το κονδύλι ε, του αντικτύπου της χρηματοδότησης. Εδώ ε, μιλάμε για κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι καν διαπιστευμένα. Χρειάζεται να παίξεις, ε, να συνεργαστείς με τοπικούς παίκτες και πίσω από αυτά τα ποσά ανέφερα, πέρσι υποστηρίξαμε με 44 εκατομμύρια τη μικροχρηματοδότηση. Ε, πρέπει να έχεις πάρα πολύ ε, μικρές εκταμιεύσεις, δηλαδή μερικές φορές 20.000 ή ακόμη και λιγότερο. Αυτά τα κονδύλια λοιπόν κατανέμονται σε ένα τεράστιο αριθμό project. Ε, υπάρχει ουσιαστικά εκταμίευση ε, των χρημάτων. Μερικές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις, μερικές φορές πρέπει να διασφαλίσεις ε, ότι ε, το άλλο μέρος έχει και την απαραίτητη κατάρτιση. Αν παραδείγματος χάρη θέλουμε μια οντότητα να κινηθεί προς τη μικραχρωμοδότηση, θα πρέπει να έχει και τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για να κινηθεί προς τα εκεί εμείς έχουμε κάποια θετικά μηνύματα. Δηλαδή φτάσαμε πέρσι κοντά στην εκταμείευση του ενός δισεκατομμυρίου. Είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δηλαδή, ε, καθυστερούμε γιατί βάζουμε και κάποιες προϋποθέσεις στα δανειά μας, κάποιους όρους, γιατί θέλουμε να δούμε αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε αν ε, τα κονδύλια που εκταμιεύουμε, ε, που κατανέμουμε, οδηγούν σε κάποια συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα. Η κυρία Για μένα το πρόβλημα είναι με αυτά που μας είπατε, που νομίζω ότι ναι, μένει, οι προθέσεις σας είναι πολύ καλές, αλλά δεν μου εξηγείτε πως ορισμένε πιστοτικές γραμμές που έχουν ανοίξει και είναι ανοιχτέ από το 2003, δεν υπάρχει κανένα είδο αποτελέσματο. Δηλαδή ήθελα να ξέρω πού οφείλεται αυτό και με ποιο τρόπο η τράπεζα αλλάζει την προσέγγισή της. Την προσέγγισή Γιατί πολύ ωραία να κάνετε αυτό το τεχνικό συμβούλιο, αλλά ίσως η τράπεζα θα πρέπει να μάθει πώς από τη μικροχρηματοδότηση εγώ είχα και πάρα πολλές ε, εμπειρίες ε, στη χώρα μου. Ε, δεν είναι λοιπόν τόσο δύσκολο να γίνει. Το πρόβλημα είναι αν είναι διαφορετική η νοοτροπία. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί να μεταχειριστεί έναν άνθρωπο που έρχεται για μικροχρηματοδότηση με τον ίδιο τρόπο που θα μεταχειριστεί στην τράπεζα Σανταντέρ. Ποια είναι λοιπόν η ειδική τεχνική που χρησιμοποιεί η τράπεζα για τη μικροχρηματοδότηση και πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Έχουμε μια σειρά υπογεγραμμένων συμβάσεων που τουλάχιστον μέχρι τώρα ε, και έχουν περάσει 14 χρόνια έτσι από το 2003 δεν βλέπω καμία έκβαση. Δηλαδή, εντάξει, δεν μεν έχετε καλέ προθέσει, αλλά να μου πείτε εδώ υπάρχει συγκεκριμένο συγκεκριμένος αριθμός συμβάσεων υπογεγραμμένων, αλλά πού είναι τα αποτελέσματα. Βλέπω εδώ 0, μηδέν. Τι συμβαίνει λοιπόν, ε, τι γίνεται στην παρασκήνη και πώς ακριβώς το σκέφτεται όλο αυτό η τράπεζα. I Ευχαριστώ για το ερώτημα και καταλαβαίνω τι ήταν Η προσέγγιση μας είναι να διασφαλίζουμε σε ό,τι αφορά την αφετήρια. Ξεκινώ λοιπόν από την αρχή. Δεν στηρίζουμε δηλαδή μόνο τι ε, ήδη παγιωμένε και δρεωμένε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θέλουμε πολύ περισσότερο να στηρίξουμε ε, τον τραπεζικό τομέα μέσω, τον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζών, οι οποίε κάνουν εξαιρετική δουλειά βέβαια, αλλά δεν ε, έχουν σχέση με ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο ε, στρέφεται προς ε, τα μικροδάνεια. Για πολλά χρόνια λοιπόν έχουμε καταλάβει, εδώ και πολύ καιρό έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να πάμε παραπέρα. Πρέπει να βρούμε ομολόγους που σίγουρα δεν θα είναι τόσο εδρεωμένοι, δεν θα έχουν δηλαδή το επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν ε, εδρεωμένοι φορείς, με δίκτυα, κεφάλαια και το καθεξής. Ισχύει ότι είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο, κάτι πολύ πιο ε, χρονοβόρο, μόνο και μόνο για να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς ε, θέλουμε από εκείνους. Και σίγουρα το ίδιο ισχύει και για τα πρότυπα, τους κανόνες και, την, και τις αναφορές. Βέβαια, ε, πρέπει και αυτοί να ανταποκριθούν αντιστοίχως και είμαστε και εμείς πολύ επιλεκτικοί σε ό,τι αφορά την επιλογή των ομολόγων. Είναι δύσκολο να ανανεώσει βάσει καλών επιδόσεων μία πίστοση, ε, όταν κάποιος ξέρει δηλαδή πολύ καλά όμως τι πρέπει να κάνει, είναι πολύ διαφορετικό αυτό από το να βρίσκεις καινούριου ομολόγους και να ξεκινάς την ίδια διαδικασία ξανά και ξανά. Γι' αυτό και υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα θέλαμε κι εμείς ε, ε, να κατανέμονται τα κονδύλια γρήγορα και αυτό θα ήταν πολύ καλό. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε απλώς ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, Αλλά είναι, πιάνει τόπο αυτός ο χρόνος και αυτή η προσπάθεια. Και αυτά τα χρήματα, εξάλλου, όταν τους δίνουμε ε, τεχνικούς συμβούλους. Για να εξολογήσουμε την ποιότητα μίας αίτησης επίστοσης από οποιοδήποτε ομόλογο, που μπορεί να μην έχει καν επαρκή λογιστικά στοιχεία πρέπει να κατανοούμε τον κλάδο και να βλέπουμε τελικά εάν βγάζει νόημα η αίτηση ή όχι. Είναι κάτι λοιπόν που απαιτεί χρόνο. Και αν δείτε τα ποσά που δίνουμε με τις μικροπιστώσεις είναι πραγματικά μηδαμινά σε σχέση με ε, τις συνήθεις πιστώσεις που δίνουμε. Είναι λοιπόν κάτι που απαιτεί χρόνο, ενέργεια, αλλά έχει αποτελέσματα, γιατί ε, φτάνει σε σημαντικά τμήματα του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές. Μπορείτε να απαντήσετε και στα υπόλοιπα ερωτήματα. Στο Μαλάουι. Μάλιστα και τη μόχλωση. Η μόχλευση αφορά τις ε, μεμονωμένες ε, λειτουργίες μας. Οι επιχειρήσεις, όταν χρηματοδοτούμε ένα έργο, φαντάζομαι εννοείται το όριο των έργων. Η μόγλευση ήταν ιδιωτικό κεφάλαιο. Ναι. Όταν παρεμβαίνουμε συνήθως διασφαλίζουμε σε περίπτωση ταμείου για παράδειγμα δεν δίνουμε πάνω από 20-25% των ε, ιδιωτικών κεφαλαίων. Άλλες φορές καταλήγουμε σε άλλα MDBs ε, θα είμαστε εμείς δηλαδή και θα είναι και άλλες τέτοιες ε, οντότητες μάλλον. και αυτό συνδέεται με και τις χαρακτηριές γραμμές που υπάρχουν. Όμως, ε, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε υπερβολικά ποσά, γιατί θέλουμε να εμπλακούν και άλλοι επενδυτές. Δηλαδή μπορεί εμεί να δώσουμε 30% το υπόλοιπο 70% να προκύψει από την αγορά. Είπατε μόχλευση 1 προ 9. Ένα ευρώ, ε, από τα 1 ευρώ 9 επενδύονται. Είναι δημόσια κονδύλια αυτά ή είναι ιδιωτικέ επενδύσεις. Αυτό ρώτησα. Μάλιστα. Σε επίπεδα χαρτοφυλακίου λοιπόν. Είναι και τα δύο στηρίζουμε ένα έργο, δεν το χρηματοδοτούμε δηλαδή κατά 100%. Τα υπόλοιπα πρέπει να προκύψουν είτε από την αγορά, είτε από ε, κρατικούς φορείς, άλλες τράπεζες. Γι' αυτό έχουμε αυτόν τον πολλαπλασιαστιακό παράγοντα, αλλά αυτό συνδέεται και με την ανακύκλωση των πόρων όταν έχουμε ε, επιστροφή δηλαδή πόρων μετά την εκταμίευση, αυτά τα χρήματα επανεπενδύονται. Αν δείτε λοιπόν τον αριθμό των εγκρίσεων, υπό το EIF νομίζω ότι περάσαμε το όριο των 6 δις. Μέχρι το 2020 νομίζω θα φτάσουμε τα 10 δις ενδεχομένως. Οπότε έχουμε υπερβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, τους πόρους ε, του EIF ακριβώς λόγω τη ανακύκλωση κονδυλίων. Και επειδή ακριβώς επιστρέφουν αυτά τα χρήματα και επανεπενδύονται σε άλλα έργα, έχουμε φτάσει και σε ένα βιώσιμο επίπεδο ε, ετησίων πιστώσεων της τάξης των 800 εκατομμυρίων, χωρίς να χρειαζόμαστε πλέον άλλους επιπρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ιδιωτικά, τα, τα κεφάλαια πόσα είναι. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι τα ε, δημόσια κονδύλια κινητοποιούν μόνο δημόσια. Ε, τα δημόσια κονδύλια στη, της ΕΤΕΠ πόσα ιδιωτικά κινητοποιούν. Δεν έχω ακριβή αριθμητικά στοιχεία, αλλά για να σα δώσω μια πρώτη αντίδραση. Από αυτό το πολυπλασιαστικό παράγοντα, ένα, τον λόγο δηλαδή 1 προ 9, λέει κάτω από το μισό αφορά την ε, επαναχρησιμοποίηση ε, των πόρων. Οπότε τι υπόλοιπε φορές ε, σίγουρα πρόκειται για τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα τη χρήση αυτών των πόρων. Δηλαδή μέχρι τα 5 το λόγο του 5, 1 προς 5 είναι επειδή δίνουμε εμείς ένα σημαντικό ποσό και το υπόλοιπο προκύπτει από το γεγονός ότι επανεπενδύουμε ε, και συμπληρώνουμε το χαρτοφυλάκιο με νέες επιχειρήσεις. Αυτά εν ενδεικτικών στοιχείων. Ωραία. Στείλτε μας και μία επιστολή για να μας δώσετε συγκεκριμένα νούμερα. Και ευχαριστούμε εκ των προτέρων και για ε, όσα μας είπατε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Για το Μαλάουι και την αποθήκη γεωργικών προϊόντων είναι ένα έργο με την τράπεζα στο Μαλάουι, αλλά είναι αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα το έργο αυτό. Εμείς εξετάζουμε κάθε χορήγηση κονδυλίων, αυτό το εξετάζουν οι ειδικοί μας από το γεωργικό τμήμα. Είναι ε, μία δράση για να δώσει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα και να εξετάσει κάθε ε, δράση χωριστά και συμπληρώνει ένα κενό που υπάρχει όχι μόνο στο Μαλάουι αλλά και σε πολλά άλλα μέρη. Είχαμε αιτήματα και από άλλες χώρες ΑΚΕ για να κάνουμε κάτι παρόμοιο στις χώρες τους γιατί χάνονται πολλά χρήματα από την απώλεια της σοδιάς. Και ε, έτσι η αξιακή αλυσίδα μετά την ε, σοδία ε, προστατεύεται. Καλή επιτυχία, γιατί ειδικά στο Μαλάουι είναι παλιό το θέμα και απέτυχε το έργο γιατί αυτοί που υλοποιούσαν το έργο δεν ήθελαν να δωροδοκίσουν τη διεφθαρμένη κυβέρνηση εκεί και γι' αυτό αποσύρθηκαν. Το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες χώρες. Η, ε, το πρόβλημα της ε, Αφρικής είναι ότι δεν μπορούν να αποθηκεύουν την ε, πλεονάζουσα γεωργική εσοδεία. Και μετά αυτό, μεταξύ άλλων, προκαλεί και λοιμό. Να ρωτήσω κάτι τη βιωσιμότητα των έργων, πώς την παρακολουθείτε. Δηλαδή, αν ολοκληρώθηκε ένα έργο πριν από πέντε χρόνια. Γίνεται συστηματική παρακολούθηση για να δείτε τι απέγινε από αυτό μετά από μια πενταετία. Ή απλώς ελπίζουμε το καλύτερο από μακριά. Η κυρία Κάπελ. Τελευταία συμπληρωματική ερώτηση δεν έχουμε χρόνο. Ακούσαμε ότι το 2016 αυξήθηκαν οι δαπάνες κατά 63% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό πώς εξηγείται. Και δώστε μας και ένα παράδειγμα, με πού πήγαν, πού διοχετεύθηκαν τα κονδύλια αυτά. Για την παρακολούθηση πριν ε, συμμετάσχουμε σε ένα έργο θα υπάρξει δέουσα επιμέλεια. Υπάρχει λοιπόν ε, μια ομάδα που ε, διασφαλίζει ότι το έργο αυτό έχει όλα τα στοιχεία, έχει την αξία του και τα κονδύλια διοχετεύονται συγκεκριμένα στην υλοποίηση του έργου, του συγκεκριμένου δηλαδή. Η παρακολούθηση γίνεται συστηματικά γιατί προκύπτει από τις συμβάσεις μας. Ε, έχουμε δηλαδή, το δικαίωμα ε, να ζητούμε πληροφορίες, να επισκεπτόμαστε ε, τις εγκαταστάσεις και ανέφερα προηγουμένως και τη διαχείριση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, που είναι σαν ένας πίνακας επιδόσεων και εκτιμούμε ένα έργο ακριβώς ε, με αυτό που προσδοκούμε ως ε, αντίκτυπο του έργου. Αυτό το ελέγχουμε και μετά την υλοποίηση σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Και αυτό το ε, συζητούμε με τον ομόλογό μας. Σίγουρα το προκολουθούμε αυτό. Ετησίως εκπονούμε και ένα έγγραφο που κάνει μια επισκόπηση ε, της κατάστασης και ο πίνακας επιδόσεων επίσης επικαιροποιείται. Δεν είναι δηλαδή ε, κάτι το στατικό, εξελίσσεται βάσει των ε, έργων και βάσει των διδαγμάτων που αντλούμε κάθε χρόνο. Για την εκταμείευση, να δώσω το λόγο στη συναδελφό μου. Ευχαριστώ. Παρακολουθούμε λοιπόν ε, τα αποτελέσματα τουλάχιστον έως και τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ε, κάποιες φορές ακόμα και αργότερα η ομάδα αξιολόγησή μας θα επιστρέψει για να εξετάσει τις, ε, τα αποτελέσματα ενός έργου. Για μας είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την μακροχρόνια λοιπόν, παρακολούθηση ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Για τις εκταμιεύσεις θα ήθελα λίγο ε, να σας πω κάτι το οποίο εξηγεί λίγο και την προσαρμογή μας ό,τι φορά την ε, οικονομική διαμεσολάβηση. Οτιδήποτε συνδέεται δηλαδή με την πρόσβαση των μικρομεσών επιχειρήσεων στις πιστώσεις είναι ότι πράγματι θέλαμε να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο και αυτό συμβαίνει βέβαια μόνο όταν τα χρήματα φτάνουν στον τελικό δικαιούχο. Γι' αυτό και το προσωπικό μας από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όταν ε, εκτιμούν μια νέα γραμμή προπολογισμού, γραμμή επίστασης μάλλον, ε, με ένα νέο ε, ενδιάμεσο, θέλουν να το βρουν από την αρχή όταν ε, το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, ε, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι η πρώτη εκταμείευση θα είναι διαθέσιμη όταν χρειαστεί. Κάποιες φορές είναι διαθέσιμη εκταμείευση κατά τη, διά... κατά τη στιγμή της υπογραφής ή το αργότερο ένα χρόνο αργότερα. Και αν δείτε λοιπόν τι συμβαίνει, θα δείτε μια σημαντική αύξηση ε, των εκταμιεύσεων που πετύχαμε τα τελευταία δύο χρόνια και αυτή είναι μια τάση που θα συνεχιστεί. Οπότε, καμία γραμμή πίστοσης δεν υπογράφεται εάν δεν είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ε, θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα, φτάσει τελικά, ε, θα φτάσουν τα κονδύλια στους τελικούς δικαιούχους και μάλιστα αλλιάν συντόμους. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ή η εισηγήτρια. Νομίζω όλα τα είπαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις ε, εξηγήσεις που μας έδωσαν και ε, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε καλή συνεργασία και στο μέλλον. Θα έχουμε και διευκρινήσεις γραπτός για το τι κάνει η τράπεζα σε συνεργασία με την Κομισιόν. Α, με συγχωρείτε, η Κομισιόν. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Τα επενδυτικά μέσα είναι σημαντικό εργαλείο για τις επενδύσεις της χώρας ΑΚΕ. Η Κομισιόν η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο, θέλει να συνεργαστεί στενά με την ΕΤΕΠ για να ε, είναι σίγουροι ότι θα υπάρχουν ε, θα υπάρχει συμπεριματικότητα και στρατηγικές που θα συνάδουν με τις ε, δράσεις μας κατόπιν ε, της σύσταση της ενδιάμεση αξιολόγηση ε, του επενδυτικού μέσου το 2010 συνεχίζονται οι προσπάθειες για να προωθήσουμε την συμπληρωματικότητα μεταξύ των project που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕΠ και την Κομισιόν. Η Κομισιόν ενθαρρύνει την ΕΤΕΠ ε, να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να προωθήσει την παρακολούθηση των επιχειρήσεων και τον ε, αναπτυξιακό αντίκτυπο του μέσου επενδύσεων σύμφωνα και με τις συστάσεις ε, της ομάδας πολιτικής ε, της πλατφόρμας για το blending. Επίσης, θα την ΕΤΕΠ να συνεχίσει τις προσπαθίες της για να αυξήσει την προσθετικότητα στις επιχειρήσεις της, να προωθήσει τη χρήση των εργαλείων ε, κεφαλαϊκού κινδύνου ε, προκειμένου να προωθήσει την ε, ιδιωτική χρηματοδότηση σε επίπεδο προγράμματος οι κατευθυντήριες γραμμές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 συμφωνήθηκαν με την ΕΤΕΠ οι επιχειρήσεις είναι μία από τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος ε, της ευρωπαϊκής βοήθειας. Εμείς καλωσορίζουμε την αύξηση της εκταμιεύσεις ε, και ε, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των επενδύσεων της ΕΕΠ. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων, αυτό έχει προσαρμοστεί από την Κομισιόν και θέλουμε να έχουμε περαιτέρω δραστηριότητες blending για να έχουμε μόχλευση 44 δισεκατομμυρίων στην Αφρική και στην γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Ο στόχος ε, αυτού του σχεδίου είναι διτός ε, να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να καταπολεμήσει κάποιες από τις αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης. Ε, ε, έχουμε και μία ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες των εταίρων μας. Έχουμε ε, συμμετοχή στο Στρατηγικό Συμβούλιο της ΕΤΕΠ. Αυτό φυσικά θα συνεισφέρει και στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε και αυτό το σημείο. Το θέμα της συνεργασίας θα το δούμε χωριστά να ενημερωθούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε για την παρουσίαση και πάμε στο τελευταίο σημείο. Το σημείο 15 που είναι η εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Στη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Ο κύριος Πούφαν είναι από το ελεγκτικό συνέδριο αρμόδιος για αυτό το θέμα και θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεση αυτή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μας η προστασία της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα και την προσβασιμότητα του νερού ήταν ένα στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά έτη. Θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των καταναλωτών, να, καταπολεμήσουμε τις αρνητικές ε, συνέπειες ε, μόλυσης του νερού. Η οδηγία για το πόσιμο νερό θέτει τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, για την ανθρώπινη κατανάλωση. Η οδηγία ζητά από τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν μία έκθεση για την επικαιροποίηση της κατάστασης του νερού που προβλέπεται για ανθρώπινη κατανάλωση κάθε τρία έτη. Μια άλλη επικαιροποιημένη ενημέρωση για την ποιότητα του πόσιμου νερού θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη για τον καταναλωτή. Ο έλεγχος μας επικεντρώθηκε στην οδηγία του πόσιμου νερού και εξετάσαμε αν έγιναν σεβαστές ε, οι απαιτήσει και αν ένας ε, αριθμός έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο συνοχή και τα Περιφερειακά Ταμεία Συνοχής βελτίωσαν την ποιότητα του πόσιμου νερού και την καλύτερη πρόσβαση σε αυτό. Εξετάσαμε αν ε, η ροή της χρηματοδότησης ήταν επαρκής για να εγγυηθούμε την βιωσιμότητα ε, των ε, υποδομών διανομής πόσιμου νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε τον έλεγχό μα, επικεντρωνόμενοι στα κράτη-μέλη που ε, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και μετά. Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία ήταν οι χώρες που επιλέχθηκαν ως ε, τα τρία κράτη-μέλη που ε, ουσιαστικά συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% των ε, κονδυλίων που εκταμιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν μετά το 2004. Διαπιστώσαμε ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η Κομισιόν παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς ε, τη διαδικασία σύμφωνα με την οδηγία και από το 2016 την εθνική νομοθεσία ε, για το αν ήταν σύμφωνοι με όλες τις απαιτήσει. Παρ' όλα αυτά, εντοπίσαμε μία σα κενών ε, σε αυτή την παρακολούθηση στα τρία κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε. Βρήκαμε ότι όλες οι επετόμενες παράμετροι δεν ε, επιβλέπονται. Αυτό ισχύει και για ένα project που εξετάσαμε. Είδαμε ότι τα κράτη-μέλη καθυστερούν να ε, κοινοποιήσουν στοιχεία για την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας. Ε, τα ε, κράτη-μέλη καθυστερούν να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες ό,τι αφορά την ανθρώπινη κατανάλωση. Στα τρία κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε, είχε μεταφερθεί σωστά στην εθνική νομοθεσία αυτή η απέτηση, όμως ε, είχαμε σημαντικές ε, διαφοροποιήσεις ε, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των πληροφοριών στους πολίτες. Και επίσης οι μετρήσεις για την ποιότητα του νερού δεν διατίθεται συστηματικά στους πολίτες. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει ε, να σεβαστούν την οδηγία για το πόσιμο νερό και πρέπει να αντιμετωπίσουν υψηλά ποσοστά απώλειας νερού. Είδαμε μεγάλες απώλειες ε, λόγω κακής συντήρησης των δικτύων διανομής που χρειάζονται να ε, ανακατασκευαστούν. Είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό απώλειας ε, στα δίκτυα ίδρυυση ε, και σε ορισμένε περιπτώσεις οι απώλειες έφταναν στο 60%. Θα πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους ε, για να έχουμε τις κατάλληλες επενδύσεις και να διατηρείται η ποιότητα των υποδομών χάρη στις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά τα κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια των κονδυλίων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2007-2013 θα επενδύσουν ακόμα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες οι απαραίτητες επενδύσεις ε, θα υλοποιηθούν ιδίω στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά μας έχουμε εκδώσει πολλές συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι μια, ένας πολύ σημαντικός έλεγχος που δεν αφορά μόνο τα ε, αριθμητικά στοιχεία, αλλά έχει ως ε, σκοπό να εντοπίσει τις αδυναμίες ε, στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και συνεχίζω στα γερμανικά. Ο εισηγητής έπρεπε να πάει να ψηφίσει σε άλλη επιτροπή. Με εξουσιοδότησε λοιπόν να σας ευχαριστήσω ήταν ασυνήθιστος αυτός ο έλεγχος που αφορά τις διατάξεις της οδηγίας για το νερό. Να διαβάσω τις συστάσεις του εισηγητή τώρα. Καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος από την Κομισιόν παράλληλα με τις διατάξεις της οδηγίας. Καλύτερη ενημέρωση. Δυστυχώς δεν μπορούν να αναγκαστούν τα κράτη ε, μέσα από, ε, να, να ε, παρουσιάζουν έκθεση για μικρές ζώνες νερού, αλλά και οι μικρές πρέπει να εξεταστούν και να συμπεριληφθούν γιατί συνιστούν κινδύνους. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, Υπάρχει αντιμόνιο, ε, υδράργυρος, βενζόλιο. Έχουν ανοιχνευθεί αυτά στο νερό. Βιωσιμότητα των υποδομών ο, είναι σημαντική για τον ε, εισηγητή και η συμμετοχή των πολιτών στη διατήρηση της υποδομής να μην πληρώνει το λογαριασμό μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκείνοι που ωφελούνται από τις δομές αυτές. Και ο στόχος μας θα είναι να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από ε, το εισόδημα. Οι συστάσεις ε, του οσηγητή προσανατολίζονται προς τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Ερώτηση στην Επιτροπή γιατί δεν ε, καλύπτονται και οι μικρές ζώνες παροχής νερού. Το χρονικό περιθώριο των 30 μηνών, το, το, η, χρονική καθυστέρηση των 30 μηνών που οφείλεται και η, οικονομική υποστήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης η δημοσιονομική στήριξη από τον ενωσιακό προϋπολογισμό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση από τον εθνικό προϋπολογισμό. Πρέπει να εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία η Κομισιόν και μετά το ελεκτικό συνέδριο, κυρίως Βάκενχουτ, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την σημερινή συζήτηση. Πριν ε, επισέλθω στα ερωτήματά σα Να κάνω κάποια γενικά σχόλια πρώτα για την έκθεση. Να επισημάνω ότι από δική μας, ε, τη δική μα άποψη είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην εφαρμογή τη ε, οδηγία για το πόσιμο νερό που έχουν αναγνωριστεί και από το δικαστήριο, όπως υψηλή ποιότητα πόσιμο νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και η άμεση μεταφορά ε, τη οδηγία στι τρει χώρε που έτυχαν εξέταση και μελέτε. Υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία που, έχουν, που έχει εντοπίσει το ελεγκτικό συνέδριο ε, σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των ελέγχων, διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικέ εθνικέ πρακτικέ σε ό,τι αφορά την ε, ενημέρωση του κοινού και αυτό ε, βέβαια εντάσσεται στι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Επίσης, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν και άλλες ε, ανεπάρκειες και λήψεις, όπως οι απώλειες ε, υδάτων, το θέμα των ε, μικρών δικτύων, μικρών παροχών νερού, που αναφέρατε και κύριε Πρόεδρε, η ενημέρωση του καταναλωτή, και αυτά υπάγονται στο σημερινό πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για το πόσιμο νερό. Όμως, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου τα επικαιροποιημένα στοιχεία τα εξετάζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μπει σε μια πολύ εμπεριστατωμένη διαδικασία αναθεώρησης γιατί ξέρετε ότι η οδηγία για το Πόσο νερό θα ενταχθεί σε μια νέα πρόταση που θα υιοθετηθεί πριν τα τέλη της χρονιάς. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν του 2017 και έτσι πρέπει να πω και να επισημάνω και να με ιδιαίτερη έμφαση ότι είναι πολύ επίκαιρη η ε, έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Συνδέεται με, ε, με πολλές από τις εργασίες μας και έχει αποτελέσει έμπνευση για το έργο μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και για τις πολύ σωστές συστάσεις που κάνατε. Στην αξιολόγηση δικτύπου που ε, συμπληρώνει και αποτελεί το θεμέλιο της νέας πρότασης που θα υποβληθεί σύντομα, Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχουμε δανειστεί, που έχουμε αντλήσει δηλαδή από την έκθεση για να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Τώρα, για επιμέρου θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, αλλά σίγουρα μα ενδιαφέρουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας ε, για το νερό. Η οδηγία πλαίσιο για το νερό ε, ζητά τη θέσπιση πρακτικών ε, για την αύξηση της ε, αποδοτικότητας ε, και της καλύτερης χρήσης των υδάτινων πόρων και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το ΕΣΥΦ θα εξεκολουθεί το θα εξακολουθεί να στηρίζει αυτή την εφαρμογή και θα διερευνήσει και θα αξιοποιήσει ότι ε, μέσο είναι διαθέσιμο, ιδίω για, για τον περιορισμό των απολειών υδάτων. Τώρα, να σχολιάσω τα ερωτήματά σας και να δώσω απαντήσεις. Το πρώτο ερώτημα αφορά την ε, μη υποβολή αναφορών για τις ε, μικρές ζώνες παροχής ε, ύδατος. Δεν προβλέπεται από την οδηγία αυτή τη στιγμή στις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών. Προβλέπεται αυτή η υποχρέωση μόνο για τις μεγάλες ζώνες. Προφανώς, οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την γενική συμμόρφωση σαφώ και ισχύουν και για αυτές τις μικρέ ζώνε, αλλά απλώ όχι υποβολή αναφορών. Τώρα, στη διαδικασία αναθεώρησης εξετάζουμε γενικώ τι ε, υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και θέλουμε να έχουμε και πιο ε, έγκαιρες και στοχοθετημένες αναφορές να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες για να υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία που είναι πολύ σημαντικό θέμα για τους ε, πολίτες και το αναφέρατε και εσείς κυρία Πρόεδρε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερο τους πολίτες γιατί συνδέεται στενά με την υγεία και πρέπει και εμεί να κάνουμε κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά την διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφορία για να διασκεδάζουμε τι ανησυχίε των πολιτών και να του επιτρέπουμε να έχουν μια πολύ καλή εικόνα τη ε, κατάσταση ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ενισχυθεί κατά τη διαδικασία, κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης, μαζί με περισσότερες διατάξεις για τη διαφάνεια γενικότερα. Σε αυτή την οδηγία πρέπει να δούμε και το θέμα της απώλειας υδάτενων πόρων ε, υπό το πρίσμα της διαφάνειας στις χώρες που βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση των, της απώλειας υδατινών πόρων, αυτέ, αυτό ε, δημιουργεί πιέσεις προς τις ε, εθνικές αρχές ε, να αναλάβουν μέτρα και δράση. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι αυτά είναι θέματα επικουρικότητας και γι' αυτό υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τώρα, για τι ε, καθυστερήσει ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση εκθέσεων για την ποιότητα του πόσιμου νερού που θίξατε κυρία Πρόεδρε, εδώ αναγνωρίζουμε ότι το σύστημα υποβολή αναφορών που προβλέπεται από την οδηγία σημαίνει ότι εμείς ε, δημοσιοποιούμε μία ε, παροχημένη ουσιαστικά έκθεση που παραπέμπει σε στοιχεία τριετίας. Αυτό σίγουρα δεν μας ικανοποιεί και σαφώς και εξετάζουμε τρόπους βελτίωσης αυτής της κατάστασης η καλύτερη λύση είναι να δούμε τις τεχνολογίες, τις σύγχρονες τεχνολογίες που θα μας επιτρέπει ε, να έχουμε άμεση τροφοδότηση στοιχείων δηλαδή. Και κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική αυτή συμβολή και να ε, επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο βαθμό του δυνατού προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις ε, στα όσα θα κάνουμε στην αναθεώρηση της οδηγίας. Ε, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί ε, το Σώμα των Επιτρόπων δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί, αλλά σίγουρα το σύνολο των συστάσεων έχουν τροφοδοτήσει την διαδικασία αναζήτησης και αναθεώρηση της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είσαστε πολύ πιστικός. Λυπάμαι διότι οι συνάδελφοι από τις χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία δεν τα άκουσαν όλα αυτά και δεν έλαβαν υπόψη τους την έκθεση που είναι ορόσημο εις ό,τι αφορά το τι μπορεί κανείς να κάνει για τον πληθυσμό. Κρίμα και πάλι κρίμα. Που ενώ τους αφορά δεν θεωρούν ότι έπρεπε να είναι εδώ. Λοιπόν, το ελεγκτικό συνέδριο. Μιλήσατε για την Ουγγαρία και τις πολύ ακριβές υπηρεσίες κατά 26% παραπάνω. Και πώς εξηγείται αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοούμε πάρα πολύ καλά τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής. Γενικά σε όλες τις χώρες που κάναμε τον έλεγχο μιλάμε για μικρά ή για μεγάλα project. Ξέρω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Κάτι πιο σημαντικό έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτών, γιατί οι πολίτες είναι οι δικαιούχοι αυτού όλου του έργου για την ποιότητα του νερού, αυτοί είναι που υποφελούνται. Και έχουμε πολύ καλούς ε, πληροφορικούς για να φτιάξουν ένα σύστημα λογισμικού, έτσι ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο με διαφάνεια. Αυτό για κάθε περιοχή όπου κάνουμε έργα και να βελτιώσουμε και τη συνεργασία και την επικοινωνία με την Κομισιόν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Πράγματι, κάναμε τον έλεγχο και στην Ουγγαρία. Είναι μια χώρα που και αυτή έχει κάποια προβλήματα. Ίσως ε, η επικοινωνία μεταξύ των ελεγκών, των ελεγκτών και των ε, Ουγγρικών Αρχών να μην ήταν καλύτερη, όμως την επόμενη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε καλύτερα. Μάλιστα. Στην Ρουμανία οι καθυστερήσεις και η ακρίβεια στην Ουγγαρία. Γι' αυτά τι έχετε να πείτε. Οι ακριβές υπηρεσίες στην Ουγγαρία και οι καθυστερήσεις στην Ρουμανία. Υπάρχουν κάποιες περιοχές ε, με project που είναι υποκαθυστέρηση. Μιλώ για τη Ρουμανία, γιατί είναι η χώρα μου και την ξέρω πολύ καλά. Πριν ε, κάποιους μήνες είχαμε μια νέα κυβέρνηση, έχουν αλλάξει οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς. Έτσι λοιπόν έχει χάθει κάποιος χρόνος. Κοιτάξτε, όλα τα έργα για την ε, ίδρευση είναι πολύ σημαντικά για οποιοδήποτε πολιτικό ο οποίος ε, ε, αν θέλει να επανεκλεγεί την επόμενη φορά, πρέπει να κάνει κάτι για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε την απόσταση μεταξύ υπαίθρου και πόλεων γιατί διαφορετικά μένει πίσω η ανάπτυξη της χώρας. Äh, Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα, κοιτάζοντας ποια είναι η κατάσταση στις άλλες χώρες μέλη. Θα συναντηθούμε πάλι στις 19 Οκτωβρίου, 9 το πρωί στις Βρυξέλλες και στις 26 έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση 9 με 12 παρατέταρτο ακρόαση τεσσάρων υποψηφίων για το ελεκτικό συνέδριο. Και το βράδυ είναι ο εορτασμός των 40 ετών του ελεκτικού συνεδρίου και θα βρεθούμε και εκεί. Ευχαριστώ λίγη τη συνεδρίαση.